Καλημέρα σας κύριοι συνάδελφοι. Σας ενημερώνω σχετικά με την έκβαση της ε, χθεσινής ε, συνεδριάσεως των συντονιστών όπου χρειάστηκε περισσότερος χρόνος από ό,τι προβλέπαμε αλλά μπορέσαμε να εξαντλήσουμε την ημερήσια διάταξη την οποία είχαμε καθορίσει. Όσον αφορά την κατανομή των εκθέσεων να έχετε υπόψη σας ότι εργαστήκαμε πολύ σκληρά οπότε ε, αποφασίσαμε ε, να, να βάλουμε ορισμένες αποφάσεις ε, μεταξύ συντονιστών διότι συμφωνήσαμε ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή ημέρα ε, για να μπορέσουμε ε, να ξανασυζητήσουμε ε, την κατανομή των εκθέσεων. Αν ως την επόμενη συνεδρίαση δεν υπάρξει συμφωνία, τότε η Προεδρία θα αναλάβει βάσει της μεθόδου Hont να κατανείμει τις εκθέσεις της διάφορες ε, πολιτικές ομάδες. Τώρα όσον αφορά τις, ε, τις μη πολιτικές αναφορές για να μειώσουμε την, το φόρτο εργασία μας το θέμα αυτό επίσης ε, αναβλήθηκε στην επόμενη ημέρα ε, ε, συνεδρίαση των συντονιστών και όσον αφορά τους ευαίσθητους χρόνους να ξέρετε ότι οι συντονιστές απεφάσισαν εχθές κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως των συντονιστών να χρησιμοποιήσουν σαν βαντεμέκουμ το έγγραφο της Προεδρίας και ε, θα σας κατανεμηθεί το έγγραφο αυτό ακριβώς για να γνωρίζετε ποιοι θα είναι οι κανόνες που θα διέπουν εις το μέλλον την ε, κατανομή μίας ε, αναφοράς και το χαρακτηρισμό της ως επίγουσας ή μερικός επίγουσας. Επίσης, ε, ε, ε, δόθη ένα γραπτό κείμενο στην Προεδρία το οποίο συγκεντρώνει τα στοιχεία της συμφωνίας βάσει της διαδικασίας η οποία απεφασίστη εάν Ε, χρειάζεται να συζητήσουμε ε, μία αναφορά η οποία έχει θεωρηθεί ως ε, τετελεσμένη. Επίσης, αν δεν έχει μοιραστεί αυτό το έγγραφο ακόμη να γνωρίζετε ότι θα σας δοθεί αλλά γενικώ θα ήθελα να σας πω ότι η συμφωνία μεταξύ των διαφόρων συντονιστών προβλέπει ότι αν υπάρχουν νέα θέματα, τα νέα στοιχεία τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα και ε, που έχει οδηγηθεί στο κλείσιμο της ε, διαδικασίας ο συντονιστής, οι συντονιστές μπορούν να λάβουν την απόφαση να ξανανοίξουν ένα θέμα που θεωρείται τελεσμένο. Αυτό απεφασίστηκε χθε στην μακρά συνεδρίαση των συντονιστών. Άλλωστε, όλοι οι συντονιστές ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο ενός ε, ο μηνύματος που είχε σταλεί στο μέσο της εβδομάδος από το ρουμανικό, ρουμανικό τύπο και περιμένουμε την απόφαση του Προέδρου Μπούζεκ. Αλλά οι συντονιστές ε, με μεγάλο ζήλο αποφάσισαν ε, ότι ε, το έγγραφο των ε, συνδικάτων της Ρουμανίας θα περιελάμβαναν τα στοιχεία τα οποία ανέφερα και ε, γι' αυτό θα έπρεπε ομόφωνα, να, ομόφωνα απεφάσισαν ε, να ξανανοίξουν αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω τον αριθμό της αναφοράς, αλλά πρόκειται για την ε, αναφορά σχετικά με την ελευθερία του τύπου στη Ρουμανία, που ήταν το τελευταίο θέμα που είχε συζητηθεί. Και ο συνάδελφός μας Ντουρκάης ε, είχε ζητήσει να έχει ένα γραπτό κείμενο ε, σχετικά με το σημείο 5 και όσο αναφορά το θέμα 6 για τις επισκέψεις ζήτησε ένα γραπτό κείμενο στο οποίο η γραμματεία ε, να ενημερώνει για, τις, ε, για ε, το πώς θα καθορίσουμε τον αριθμό των μελών που θα προέρχονται από κάθε χώρα και πώς θα κατανεμηθούν οι συμμετοχές στις αποστολές και στις επισκέψεις. Ε, ε, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ε, ζητηθούν βάσει γραπτού κειμένου στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών σχετικά με ορισμένες αμφιβολίες που είχαν οι συνάδελφοι. Και όλα αυτά έχουν αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση. Άουκεν. Πρώτα-πρώτα ήθελα να σας πω ότι δεν συμφωνήσαμε όσον αφορά το ποιος θα παρευθεί την έκθεση. Δεν συμφωνήσαμε, γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι ορθή η εφαρμογή, η ερμηνεία του συστήματος DEONT όσον αφορά ε, το, το ποιος θα χρεωθεί αυτή την ε, έκθεση. Επομένως, θα πρέπει να αποφύγουμε να λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις αφού διαφωνούμε. Άρα θα πρέπει να δούμε επίσης τώρα πώς θα γίνει η οργάνωση των αποστολών των επισκέψεων. Θα πρέπει να έχουμε μια γενική έποψη. Και τελικά αυτές οι αποστολές, οι ερευνητικές, ε, αυτές είναι η ε, ε, πιο σημαντική αποστολή μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή εχθές είχαμε μία περίπλοκη συνεδρίαση των συντονιστών, ότι ε, καταρχήν τα θέματα συμφωνήθηκε να συζητηθούν εις τους συντονιστές και επειδή ε, δεν παρουσιάστηκε ε, πολύ σαφώς αυτό που είπαμε χθες είπαμε ότι η καλύτερη λύση είναι ε, να συνέλθουν οι συντονιστές και να βρουν ένα σωστό τύπο πώς θα προχωρήσουμε. Βέβαια η πρόεδρος προσπάθησε βάσει του συστήματος DeHont να κάνει μια κατανομή των εκθέσεων αλλά δεν τα κατάφερε και γι' αυτό είπαμε ότι στην επόμενη ε, συνδρίαση θα βρούμε μία λύση και άπαξ και θα έχουμε ένα σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα και όλα θα πηγαίνουν καλά. Άρα θα αφήσουμε ακόμη σε κρεμότητα τα θέματα τα οποία είναι προς συζήτηση κατά τρόπον ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να έχει μία, ένα σαφές κείμενο ε, και τρόπο εργασίας. Η κυρία ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με τον μηχανισμό της συνεργασίας ακριβώς όπως το επεσήμαναν οι συντονιστές και όπως ε, επίσης είπαμε θα πρέπει να συζητήσουμε και για τα της ελευθερίας του τύπου στην Ρουμανία. Το Δεκέμβριο τα συζητήσαμε, ήρθα σε επαφή με τον ε, σύμβουλο τον ακόλουθο ε, της ε, Ρουμανίας και η λύση η οποία τελικά δόθηκε ήταν μια νίκη και αυτό δείχνει το πόσο, πόσο είμαστε αφοσιωμένοι στη, στο να δίνουμε αγώνα για τις ε, ελευθερίες, για την προστασία του πολίτη. Επομένως δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε αυτή την νίκη που όπως Τελικά εδώ πέρα διαμορφώθηκε στις ε, στις, στη, στην Επιτροπή μας μια συνένεση, επομένως ε, πρόκειται τελικά για μια νίκη κατά της ε, αυθαιρεσίας. Επίσης δόθηκε διέξοδο στο αδιέξοδο που υπήρχε προηγουμένως. Βρεθήκαμε μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά πάντως νομίζω ότι πάρα πολύ αγαστή ήταν η συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων. Οι συντονιστές χθε το απόγευμα ε, συμφώνησαν σε κάτι σαν μνημόνιο, memorandum, ε, ούτως ώστε ε, κάποιες αναφορές να εξετάζονται κάπως σαν κατεπήγοντα. Άρα θα μπορούν να ανοίξουν τις αναφορές και οι συντονιστές. Σήμερα επομένως, ό,τι χρειάζεται το έχουμε στα χέρια μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου κρίσει τέτοιου προβλήματα στο μέλλον. Νομίζω ότι πρόκειται για μια επιτυχία για μα για την Επιτροπή μα. Επίση πρέπει να σα τονίσω το ότι είμαι πεπισμένο ότι αντλήσαμε κάποια χρήσιμα συμπράσματα και μαθήματα τη Δευτέρα Δεκεμβρίου. Οπότε και εμείς ε, ω Επιτροπή τώρα έχουμε αυξημένη αξιοπιστία, έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ε, ε, δυνάμεις μας και νομίζω ότι τώρα επομένως μπορούμε καλύτερα να επιτελούμε το έργο μας δηλαδή να προστατεύουμε τον πολίτη και για άλλη μια φορά θα σας πω μπράβο μας, μπράβο μας που συνεργαστήκαμε τόσο καλά και τα πήγαμε τόσο καλά Grazie collega Bostinaro ε, quindi a questo punto procediamo con eh, un punto che abbiamo Ευχαριστώ Momento allora sobre un tema distinto pero No sé si los coordinadores ayer eh, discutieron o... οι συντονιστές δεν ξέρω αν το συντόνισε τώρα από υπόψη μου. Πάντω, εγώ θα ήθελα να πω όσον αφορά και τα πρακτικά μα. Ότι την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο ε, είχα τη χαρά και την τιμή να προεδρεύσω τη συζητήσεω. Για την οποία η, η πρόεδρο, υπό την ιδιότητα τη εισηγητρία, παρουσίασε μία έκθεσή μας. Εκείνη η έκθεση αφορούσε μία αναφορά προερχόταν από τη Γερμανία και εκκρεμούσε πάρα πολύ καιρό. Αφορούσε δε τους ασθματικούς και αυτές τις συσκευέ εισπνοής. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό το πόσοι από την Επιτροπή μας ήσαν εκεί ε, παρόντες σε αυτή τη συζήτηση η οποία προερχόταν από εμά, από την Επιτροπή μα. Επομένω, θα πρέπει να σα πω ότι με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια η πρόεδρο ω εισηγήτρια το παρουσίασε αυτό το θέμα και επίση επήρξε συζήτηση με έντονο ενδιαφέρον παρά το ότι η οργάνωση των εργασιών ήταν πάρα πολύ περίπλοκη, μια που το ανακατέψανε αυτό, ε, το βάλανε κοντά σε άλλη έκθεση που ήταν παντελώ άσχετη. Τα είπα αυτά και τα ξαναλέω το επεσήμανα από την μέρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι τη Επιτροπή μα ότι εκείνη μα η αναφορά έφτασε εσείς στην Ολομέλεια, είδε Ολομέλεια πάρα πολύ θετικά υπεδέχθη ε, την έκθεση αλλά επίσης και τις ε, προτάσεις της ε, Προέδρου μας η οποία επαναλαμβάνω ότι πάρα πολύ ωραία το χειρίστηκε. Θα πρέπει αυτό να το ξέρουν οι αναφέροντες και αναφερόμενοι. Γιατί τα θέματα τα οποία έρχονται εδώ πέρα μπορούν να φτάσουν στην Ολομέλεια. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και συμμετοχή διαφόρων συναδέλφων. Άρα, παραλαμβάνω, μπορούμε να φέρουμε σε αίσιο πέρας μία αναφορά, να κάνει όλη τη διαδρομή. Ευχαριστώ ε, τον κύριο Μαρτίνης, ε, η κυρία Νικόλο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω την απόφαση των ε, συντονιστών σε ό,τι αφορά, αφορά την ε, επανέναξη της αναφοράς για την ε, ελευθεροτυπία στη Ρουμανία. Δυστυχώς υπάρχουν δημοκρατικές διολυστήσεις. Δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι μόνο συμβαίνει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να ανησυχήσουμε όλοι από αυτές τις δύο ληστήσεις. Χρειαζόμαστε μια πιο δημοκρατική, πιο υγιή ένωση που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαίρομαι λοιπόν για την επανεκκίνηση της διαδικασίας αυτής της αναφοράς. Και χαίρομαι και για τη συνεργασία, τη συνεργασία των διαφόρων πολιτικών ομάδων που νομίζω θα είναι υποφελής για την αναφορά. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω σαφώς στο θέμα αυτό ε, κατόπιν των παρατηρήσεων που έγιναν διότι σαν Επιτροπή Αναφορών δεν λειτουργούμε για λογαριασμό μας αλλά για τους πολίτες και μόνο εάν διακομματικά μπορέσουμε να συνεργαστούμε και θέσουμε τους, τους πολίτες στο επίκεντρο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Πιστεύω όμως ότι όσον αφορά το θέμα των φαρμάκων τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Βέβαια καλύτερα θα ήταν να ήταν πιο διακομματική συνεργασία. Θα ήθελα όμως πέραν αυτού να σας πω και να γραφτεί στα πρακτικά ότι την τελευταία φορά που μιλήσαμε ε, για την ελευθερία του τύπου ή στην Ρουμανία και τη σχετική αναφορά τότε το ΕΛΚ άλλαξε μέλη και δεν εψήφισαν αυτοί οι οποίοι είχαν εκλεγεί εδώ αλλά εθνικοί βουλευτές από τη Ρουμανία που δεν είχαν συμμετάσχει εις ε, την ε, διαδικασία και δεν είχαν το ίδιο μέλημα δηλαδή να αξιολογήσουμε θετικά μία αναφορά. Άρα πιστεύω ναι. ότι στο μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες που έχουμε χρησιμοποιήσει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν. Διότι αν δοθεί αυτή η χρειά στις εργασίες του Κοινοβουλίου στο μέλλον σε αυτή την Επιτροπή, τότε δεν πάμε καλά, διότι δεν πρέπει να κάνουμε εδώ εθνικούς, εθνικές αντιπαραθέσεις, αλλά θα πρέπει να λειτουργούμε διακομματικά προς συμφέρον των πολιτών. Αυτό αναφέρεται όσον αφορά την κατασκευή κατανομή ε, των αναφορών, τι συζητήσεις και αυτή η πολιτικοποίηση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί τον τελευταίο καιρό δεν είναι προ όφελο του Κοινοβουλίου. Αλλά χαίρομαι ότι οι συζητήσεις είναι σε καλό δρόμο και ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει να είναι λιγότερο πολιτικοποιημένε οι συζητήσεις που γίνονται για επιμέρους αναφορές και ελπίζω ότι η έκκληση που κάνετε θα γίνει δεκτή από όλους με τρόπο τίμιο και υγιή. Πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η έγκριση των πρακτικών. Όχι, έκανα λάθο Ο Βέρνερ. Με συγχωρείτε, έχω μία ερώτηση την οποία έκανα και εχθές ότι όσον αφορά την ε, νομοθεσία για, την, ε, ε, για τις ακτές στην Ισπανία και εγώ έλαβα ένα ανησυχητικό μήνυμα στο μέλλον ότι θα κρατικοποιηθούν οι αμφισβητούμενες περιουσίες ενώ ουσιαστικά ε, οι, οι κάτοικοι μπορούν να πληρώσουν και να χρησιμοποιήσουν το ακίνητο που έχουν δεσμεύσει και ελπίζω ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν πολιτικές αποφάσεις εδώ αλλά θα πρέπει να ε, ενδιαφερθούμε για το συμφέρον των ε, ε, των πολιτών και διακομματικά να μπορέσουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντά τους και τα ενδιαφέροντά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το συγγνώμη και θλίβομαι που δεν ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό και ελπίζω στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Γιατί όπως είπα και στην αρχή της συνεδρίασης συζητήσαμε μέχρι τις 7 ε, παρα 20 το θέμα της, ε, του καταμερισμού έτσι, των γνωμοδοτήσεων και των εκθέσεων. Πάντω ε, ενδιαφέρομαστε πρώτα να ασχοληθούμε με τα συμφέροντα των πολιτών και μετά με των πολιτικών ομάδων. Συμφωνώ με αυτό που είπατε και νομίζω ότι το επικύρωσαν και με τα λόγια τους και οι άλλοι ομιλητέ. Ε, στο μέλλον λοιπόν ε, θα, κάνουμε, θα δώσουμε μάχη όχι για να ακουστούν περισσότερο οι πολιτικές ομάδες αλλά για να ακουστούν περισσότερο οι φωνές των πολιτών. Ε, και εγώ σας δεσμεύομαι το προσωπικό, θα το βάλω σε επόμενες συνεδριάσεις στα πρώτα σημεία της ατζέντα. Λοιπόν, θέλω να, να εγκρίνουμε τα πρακτικά της ε, συνεδρίασης 1ης και 2 η ε, Δεκεμβρίου που, δεν που αναβάλαμε χθε. Είχαμε προβλήματα χθε, θα θυμάστε. Θεωρώ ότι λοιπόν εγκρίνονται τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, έτσι, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Πολύ ωραία. Εγκρίνονται. Όπω είπα χθε, στην έναρξη τη συνεδρίασης, Τροποποιήθηκε ελαφρά η ημερήσια διάταξη, επομένως το σημείο 13 αναβλήθηκε και θα πάμε κατευθείαν στο σημείο 14 που είναι η γνωμοδότηση για την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους. Είναι μια γνωμοδότηση η οποία δυστυχώς έχει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή μας στην επόμενη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου. Γι' αυτό, λοιπόν, ζήτησα από τη Γραμματεία να επιταχύνει τις διαδικασίες και σας ζήτησα να σας μοιράσει ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας. Και μου ζήτησαν οι συντονιστές ε, να τροποποιήσουμε ακριβώς την ατζέντα της Επιτροπής μας λόγω του ότι έχουμε αυτές τις ε, επιταγές του χρονοδιαγράμματος, αν θέλετε. Αυτά τα, αυτές τις πιέσεις του χρονοδιαγράμματος. Το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο μοιράστηκε ε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι ένα σχέδιο το οποίο Καταρχάς, θέλουμε να εκφράσουμε την ε, ικανοποίησή μας ε, για την προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα. Κάποια στοιχεία θέλω να αναφέρω. Με την παρέμβασή μας ε, στη δουλειά της Επιτροπής ΙΜΚΟ, επικεντρωνόμαστε λόγω της φύσης της Επιτροπής μας στον πολίτη και στα δικαιώματα των πολιτών και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια από τα 18 σημεία που αποτελούν αυτή τη γνωμοδότηση που πρέπει να αξιολογήσουμε. Θα πρέπει η Επιτροπή μας να υποστηρίξει ιδίω το σημείο 5, το αίτημα που διαμαρφώνουμε στο σημείο 5, όπου ζητάμε από την Επιτροπή ή μάλλον συμφωνούμε με την έκκληση της Επιτροπής προς τα κάτι μέλη να μειώσουν το έλλειμμά τους ως προς τη μεταφορά των οδηγιών της ενίας αγοράς στο εσωτερικό δίκαιο σε 0,5%. Γιατί ξέρουμε πόσα παράπονα υπάρχουν από τους πολίτες λόγω αυτού του ελλείμματος και, της μεταφο... και μετα... του ελλείμματος μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν ε, και ανισότητες ε, και έλλειψη ισοπολιτείας μεταξύ πολιτών ε, διαφορών χωρών. Το σημείο 6 επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία για το έργο της Επιτροπής μας. Επαναλαμβάνουμε με αυτό το σημείο το να μειωθούν δραστικά η, να μειωθεί δραστικά η διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάση, τις οποίες κινεί η Επιτροπή. Χθε είχαμε τέσσερις αναφορές που αφορούσαν τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι αναφορές αφορούσαν αυτό το τεράστιο χρονικό διάστημα που απαιτείται. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται σωστά τα δικαιώματα των πολιτών. Και μιλάμε για τέσσερις εισάριθμες δηλαδή ε, διαδικασίες επί παραβάση ε, που κρατάνε στο διηνικές. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο και είναι σημαντικό να το πούμε και στα πλαίσια της συζήτησης που κάνουμε για την απόφαση της Κομισιόν. Γιατί εμείς αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Έπειτα. Σωστό είναι ότι η γνωμοδότηση αναφέρει διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή κάνει διάφορες εκκλήσεις προς την ε, Κομισιόν. Να προωθήσει και να υποστηρίξει το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και με τους ίδιους τους πολίτες, με τις οργανώσεις των πολιτών, με τις, με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαφόρων συμφερόντων Αυτό είναι προτεραιότητα και περνάει πριν από οποιαδήποτε άλλη υλοποίηση, αυτή η πραγματική υλοποίηση της ενιαίας αγοράς. Νομίζω ότι έχουμε αυτό το καθήκον να αναφέρουμε αυτές τις εκκλήσεις. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Τη λάβατε την γνωμοδότηση και παρότι πρόσφατα ελπίζω να είχατε το χρόνο να τη διαβάσετε. Δεν ξέρω αν κάποιο θέλει να παρέμβει για να κάνει κάποια αξιολογική κρίση για τη γνωμοδότηση την οποία σα παρουσίασα εντάχει. Sí. Eh, Θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτω. διότι όταν έχουμε μια διαδικασία αναφορών, και αν θέλουμε έτσι να σκιαγραφίσουμε τα προβλήματά μας θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε δύο προβλήματα. Καταρχήν βλέπουμε όλο και περισσότερα ότι η νομική χρήση ε, και ε, η προάσπιση των ε, συμφερόντων των πολιτών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παραδείγματο χάρη για τι ακτές της Ισπανία και τη σχετική ε, νομοθεσία πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και πιο γενικά και επίση βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά βρισκόμαστε ή πρέπει να βρισκόμαστε σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο και το δεύτερο θέμα το οποίο έχουμε είναι ότι όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν υπάρχουν παραβιάσεις, όταν αρκεί πάρα πολύ η διαδικασία παραβιάσεως της εμπιστοσύνης και συμφωνώ σε αυτά που είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής ε, ναι με να θέλουμε την ενιαία αγορά τη θέλουμε ε, και για το εμπόριο αλλά πρέπει να στηρίξουμε στο θέμα αυτό και τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής και συμφωνώ πλήρως με τα σχόλια που έχουν παρουσιαστεί επί του θέματος αυτού. Ναταλή Μπάρκερ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθουμε, να πάμε λίγο προς τα πίσω, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ε, πράξης για την ενιαία αγορά. Θα θυμάστε ότι στην ε, ακρόασή του ο Επίτροπος Μπαγνιέ είχε τονίσει και είχε πει ότι ο πολίτης θα πρέπει να μπει στο κέντρο αυτών των προσπαθειών και θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πράξη για την ενιαία αγορά εκπονήθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων ε, με έναν οριζόντιο τρόπο. Όλες οι γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συμμετέχουν και προσπαθούν να υλοποιήσουν την ενιαία αγορά. Και ο Επίτροπος Βαμπαγνιέ εξέτασε πολύ προσεκτικά όλες τις πηγές έμπνευση, όλες τις πιθανές. Την παλιά δουλειά του παλιού Επιτρόπου Μόντι, την ε, έκθεση του Λουι ε, που εκπονήθηκε στα πλαίσια της Επιτροπής ΙΜΚΟ, το Σώμα υιοθέτησε στις 27 ε, Οκτωβρίου το σχέδιο πράξης για την ενιαία αγορά που υποβλήθηκε σε συζήτηση. Υπάρχει και ένα ειδικό, ε, ένας ειδικός ιστότοπος ε, ε, για την ενία αγορά και περιμένουμε τις συνεισφορές σας μέχρι τις 28, τις συνεισφορές γενικά, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Όλες τις συνεισφορές θα τις εξετάσουμε με σοβαρότητα και προσοχή. Ο Επίτροπος και οι υπηρεσίες του συνεργάζονται εκ του σύνικης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και παρακολουθούν τις συζητήσεις της Επιτροπής ΥΜΚΟ και τις συζητήσεις των εισηγητών για τα διάφορα κεφάλαια της πράξης για την ενιαία αγορά. Της εργασίας της κυρίας Γκανιέδη, της κυρίας, του κυρίου Μπουσόη και του κυρίου Κορέια Ντεκάμπος. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 10 Δεκεμβρίου υιοθέτησε συμπεράσματα όπου υποστηρίζει τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στην ε, πράξη για την ενιαία αγορά υπό το φως των διαφόρων συνεισφορών που θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η ΕΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και όλοι οι πολίτες, οι οποίοι θα απαντήσουν ε, στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει, ο Επίτροπος θα προβληματιστεί και θα σκεφτεί τις προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στην πράξη αυτή για την ενιαία αγορά, την οριστική που θα υιοθετηθεί το ε, την Άνοιξη με βάση τα ψηφίσματα που θα υιοθετήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, η συνεισφορά της Επιτροπής Αναφορών ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα είναι σημαντική γιατί πραγματικά λαμβάνει πολλά σχόλια και πολλές ιδέες από τους πολίτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία προτάθηκαν. Νομίζω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα. Και τώρα υπάρχουν δύο θεματάκια τα οποία θα ήθελα να διευκρινιστούν. Θα ήθελα κάτι για το σημείο υπαριθμών 8. Για το 8 λοιπόν έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες για το τι θα γίνει, τι, πώς θα κρυθεί αυτή η υπόθεση, διότι πάμε μετά στο σημείο 7 όπου ένας καταναλωτής μπορεί ο ίδιος να αν λάβει την πρωτοβουλία άσκηση κάποια ε, ομαδικής αγωγής. Άρα, θα πρέπει αυτά τα δύο να τα δούμε τα σημεία τα οποία σα είπα. Κατά τα άλλα όμω είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας μίλησα για το σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για τις ε, τροπολογίε είναι η πέμπτη, 3 η ώρα το απόγευμα. Θα συλλέξουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε το κείμενο την 1η Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Και πάμε στο επόμενο σημείο. Το σημείο 15, η συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream. Η κυρία Γκέριγκερ είναι παρούσα? Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είχα ε, αναλάβει εγώ να μιλήσω εδώ στην Επιτροπή μας και κάνω μια εισήγηση για αυτό το θέμα τον Ιούλιο πέρσι και θυμάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετήθηκε πάρα πολύ θετικά, είπε ότι καλύπτεται από τα όσα αναφέρονται στο κείμενο της Nord Stream επίσης ε, και άλλα και άλλες πέντε χώρες, Γερμανία, Ρωσία, Δανία, Φινλανδία και και άλλες χώρες ε, είπαν ότι συμφωνούν και η Κομισιόν θεώρησε ότι δεν χρειάζεται να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία και ε, ε, θεώρησε ότι είναι αποδεκτή αυτή η έκθεση των επενδυτών. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι θα υποστούν κάποιες πάρα πολύ αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Επομένως, Θέλω να ρωτήσω την ε, Επιτροπή. Αυτά που λέει το άρθρο 11 της σχετικής οδηγίας, τα φροντίζει η Κομισιόν, παρακολουθεί το αν εφαρμόζονται. Δηλαδή, είναι η Κομισιόν ικανοποιημένη από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καλύπτεται η Επιτροπή από τις ε, δημόσιες διαβουλεύσεις που ισχυρίζεται ότι ο διοργάνωσε η εταιρεία, γιατί πάρα πολλέ ε, οργανώσει και φορεί είπαν ότι είναι οίκιστα ικανοποιημένοι από την ποιότητα αυτή τη ε, ε, μελέτη αξιολόγηση. Έχουμε το Ιστονικό Ταμείο για την Φύση, την Οργάνωση για τη Φύση, το, το Πράσινο Κίνημα τη Εστονία. Όλοι αυτοί παραπονούνται και έχουν προσφύγει δέκε σε δικαστήρια στην Φινλανδία μια που η υπόθεση αυτή αφορά τα χωρικά είδατα αυτών των δύο χωρών, Εστονία και Φιλανδία και είπαν επομένω ότι είναι ατελή αυτή η μελέτη των επιπτώσεων και ότι δεν καταγράφονται όλε οι αρνητικέ για το περιβάλλον συνέπειε. Ο επομένω. Θα χρειαστεί χρόνο. Έχουμε πάντω και άλλο φορέα και άλλη οργάνωση, το WWF από την Γερμανία, που θεωρούν ότι είναι ανεπαρκής αυτή η μελέτη επιπτώσεων. Επίσης, έχουν ασκήσει πίεση στην εταιρεία. Κατάφερε αυτή η WWF να αποσπάσει 10 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά κάποια πρόγραμματα για το περιβάλλον. Το θέμα είναι όμω γιατί αλλιώς τα λέει η έκθεση. Δηλαδή γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχουν προβλήματα η έκθεση, δεν υπάρχουν και αν δεν υπήρχε λόγος, αν, αν υπήρχε αμεληταίος κίνδυνος, πώς απέσπασε όλα αυτά τα, χρήματα εναντίον του κινδύνου η WWF. Επίσης υπάρχει και άλλη μια οργάνωση που φροντίζει την ε, καθαρή Βαλτική και εκείνοι απευθύνθηκαν στην εταιρεία Υπέβαλαν κάποια ερωτήματα, δεν πήραν ποτέ απάντηση. Επομένω, ούτε αυτό είναι αποδεκτό σαν διαδικασία διαβούλευση. Τέλο. νομίζω θα πρέπει να επιφυλασσόμεθα, διότι δεν είναι άρτη αυτή η μελέτη αξιολόγηση της Nord Stream. Η Nord Stream έχει χρηματοδοτήσει έρευνες, ε, από τις οποίες έρευνες προήλθε αυτή η ανάλυση, αυτή η μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων. Πάνω από 500.000, 500 εκατομμύρια δολάρια έχουν καταβληθεί από την εταιρεία αυτή ε, για σκοπού ερευνητικού επομένω. δεν μπορεί κανεί παρά να ρωτηθεί τι γίνεται. Πώ είναι εδώ να ένα μερόληπτη αυτή η μελέτη. Επίση είχαμε και κάποιου άλλου, και κάποιου ε, αλληλεί, οι οποίοι τώρα θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα του αλληλευτικού πόρου, μια που αυτό το πρόγραμμα έχει επηρεάσει αρνητικά τι ε, δραστηριότητέ του. Και είναι αλήθεια ότι η Nord Stream δίνει χρήματα στου ψαράδες. και Πολωνία. Ψαράδες επίσης παίρνουν 5.000 ευρώ αναλυτικό σκάφος και Σουηδοί επίσης παίρνουν 30.000 ευρώ ανά για τον ίδιο λόγο. Επειδή δηλαδή έχουν οι αλληλευτικοί πόροι μετακινηθεί. Έφυγαν από εκεί που ήταν. Πήγαν σε άλλες περιοχές. Είπαμε λοιπόν, όμως από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει όλοι να έχουν του ίδιου κανόνε παιχνιδιού για την ίδια αστηριότητα. Τώρα έχουμε και κάποιου άλλου εμπλεκόμενου κάποια κράτη-μέλη που το 2009, η Λετωνία συγκεκριμένα, είχαν διατυπώσει κάποιε αμφιβολίε όσον αφορά τι συνέπειε για το περιβάλλον αυτή τη υπόθεση, είχαν θέσει κάποιε δήματα ασφάλεια, όμω είχαμε και λιθουανικέ αρχέ που επίση είχαν επιληφθεί, είχαν ανησυχήσει, είχαν θεωρήσει ότι υπάρχει εδώ ζημία για το περιβάλλον και είχαν πρόβληση σε συγκεκριμένε ε, υπολογισμού. Επομένω, έχουμε εδώ ένα σωρό επιφυλάξει όσον αφορά το Nord Stream. Τέλο πάντων, ε, κατακλείδη, νομίζω ότι η Nord Stream απαντά στους εμπλεκόμενους αυτούς που καταγγέλνουν πράγματα μόνο όταν τις ασκούν κάποια πίεση. Αυτό το θεωρεί η Κομισιόν αποδεκτό, ανοιχτό και προχωρεί δε αυτό το έργο υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε ότι είναι ένα σημαντικό έργο για τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα. Θεωρείτε έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δε ιστοσελίδες της ΕΕ ή τέλο πάντων και στις σελίδες, της, ιστοσελίδες της ε, αναφέρονται κάποιες δηλώσεις από υπαλλήλους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά δίνουν το πράσινο φω στη συνέχιση του έργου. Επομένω, για πετε μα, εσεί είστε ικανοποιημένοι από αυτή την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων όπω την υπέβαλε ενό stream, είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των ε, τελεστισών διαβουλεύσεων και τι γίνεται με όλε αυτέ τι οργανώσει, του φορεί που σα ανέφερα, τι γίνεται με όλε αυτέ τι επιφυλάξει των ε, γεωργών, των, των, των, των αλλιέων από την Πολωνία, τι γίνεται, σα καλύπτουν οι εξελίξει αυτέ, τι λέει Κομισιόν. Hey. Κομισιόν έχει την, ε, τον λόγο, παρακαλώ. Νίκα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, εδώ όντως έχουμε θέμα το οποίο εκρεμεί εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκρεμεί από το 2007 οπότε τότε και υπευλήθησαν οι αναφορές έκτοτε κάναμε δύο δημόσιες ακροάσεις Είχαμε και άλλες επαφές με τους αρμοδίους εδώ στο Κοινοβούλιο και ευθύ εξ αρχής εξηγήσαμε ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα με το θεσμικό μας ρόλο τόσο ώστε να μπορέσουμε να διεξάγουμε γενικώ αμερόληπτες, ανεξάρτητες μελέτες και για αυτό το λόγο και θα, ας εστιαστούμε τώρα σε αυτό το οποίο επί αξιότιμη βουλευτή όσον αφορά τις μελέτες οι οποίες έγιναν ποιότης και αρμοδιότης του επιτελέχοντος την μελέτη. Αυτά είναι πάντα θέματα που τραβούν την προσοχή, οπότε θα πρέπει να σας πω σχετικά με αυτό ότι ευθύ εξ αρχής, όταν άρχισε αυτή η υπόθεση του έργου Nord Stream, ευθύ εξ αρχής λέγω ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν εκδώσει σχετική απόφαση το 2006. Ή σε εκείνες τι αποφάσει υπήρχαν κατευθυντήρε γραμμέ για τα 10 έργα προτεραιότητα και εκεί είχαμε έναν μακρύ κατάλογο έργων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι θα γίνουν στο μέλλον. Ε, επί τη βάση του καταλόγου θα το Κοινοβούλιο και Συμβούλιο στην απόφαση δε εκείνη είχε οριστεί ξεκάθαρα ότι το έργο όπως πάντοτε ισχύει Παρά ότι αυτό το επαναλάβουν η απόφαση, ότι το έργο επρόκειτο να είναι ε, να, συμμορφωθεί με την περιβαλλοντική νομοθεσία και συνακόλουθα θα είχαμε και την ε, μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα, όπως μας τα λέει η, η να τελικά για αυτές τις μελέτες ε, τις σε αυτέ τι υποστήριξε οικονομικά η εταιρεία. Με αυτό είναι φυσιολογικό. Και έτσι γίνεται και με τη σχετική, το προβλέπει και σχετική οδηγία. Ότι αυτό ο οποίος ε, κάνει το έργο, εκείνο παρέχει τι πληροφορίε στι αρμόδιε αρχέ. Ότι δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει και να αποσπάσει τη σχετική έγκριση. Και γιατί αυτό, διότι όλε αυτέ οι πληροφορίε που αυτό ο οποίο εκτελεί το έργο δίνει, όλες αυτές τις πληροφορίες αναλύονται με κάποιο είδους διαβούλευση και από τις αρμόδιες αρχές που τελικά θα χορηγήσουν την έγκριση. Και επομένως αναλύονται αυτές οι αποφάσεις και τελικά πρόκειται για μια τέτοια διαδικασία που ισχύει. Προβλέπονται τέτοιου είδους διαβουλεύσεις πρώτα-πρώτα με τι αρμόδιες αρχέ και άλλη μία δημόσια με τον κόσμο. Η δε πολιτή εμπειρία μου λέει ότι πρόκειται τώρα για το πρώτο έργο για το οποίο έγινε τόσο ευρία, τόσο εκτεταμένη διαβούλευση με τον κόσμο σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Αυτό γίνεται όμως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια και αλλού. Οπότε, Όποιο ήθελε είχε όλε τι ε, πληροφορίε που χρειαζόταν. Και ευθύ εξ αρχή είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μια που εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε μια δική μα μελέτη, για αυτό το λόγο και πρόκειται να παρακολουθήσουμε, να υποπτεύσουμε αυτέ τι δραστηριότητε. Και επίση, επισήμω, τα συζητήσαμε σε κάποιο είδου θεσμικού χαρακτήρα ομάδε, όπω του εμπειρογνώμονε των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν κάποιοι επιστήμονε από όλα τα κράτη-μέλη, από του 27 και πρόκειται για κάποιου οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για μελέτε επιπτώσεων και επανειλημμένα τα συζητήσαμε για να μπορούμε να διαπιστώσουμε τι πρόοδο σημειώθηκε όσον αφορά αυτέ τι μελέτε των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών και ουδέποτε σε τέτοιε συναντήσει δεν είχαμε κάποιο είδου επίσημη διαφωνία από πλευρά κάποιου μπλεκόμενου κράτου μέλου όσον αφορά το κύρο των σχετικών στοιχείων. Κύριε Πρόεδρε, μα για ποια στοιχεία μιλάμε. Μιλάμε για κάποιο είδου ε, λεπτομερή επιστημονικά δεδομένα, γιατί για όποιον δεν το ξέρει, μιλάμε εδώ πέρα για κάποιον αγωγό που ξεκινάει από τη Ρωσία και φτάνει στη Γερμανία. 1200 χιλιόμετρα. Και διασχίζει αποκλειστέ οικονομικέ ζώνε, αλλά και χωρικά ύδατα κρατών μελών που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση άδεια και έγκριση. Επομένω, σύμφωνα με την οδηγία για τη μελέτη των, των και την συμφωνία για τι διαβουλεύσει, αυτό που κάναμε ήταν από την αρχή να εξασφαλίσουμε ότι όντω θα γίνουν οι προβλεπόμενε διαβουλεύσει και είναι αδύνατο τώρα να κάτσω και να σα επαριθμίσω το ακριβώς πόσες σελίδες γραφτήκαν για αυτές τις διαβουλεύσεις πάντως. Έχουμε κάποιο έντυπο το οποίο λεπτομερώς αναφέρει τη γερμανική μελέτη επιπτώσεων. Έτσι σας το λέω αυτό ενδεικτικά. Ε, είχαμε τέτοιες μελέτες επιπτώσεων που γίνανε χωριστά στο καθένα από τα μπλεκόμενα Φιλανδία, δηλαδή Δανία, Γερμανία, Σουηδία, αλλά και στη Ρωσία και μόνο για τη Γερμανία είχαμε μια τεχνική έκθεση άνω των χιλίων σελίδων. Υπήρχε και μια σύνοψη που θα ήταν ανοιχτή στο κοινό, 48 σελίδων, εκλαϊκευμένη κατά κάποιο τρόπο, αλλά είχαμε και κάποια ειδική έκθεση όσον αφορά την προστασία της φύσης. Και είχαμε και άλλη μια έκθεση που έγινε αιτήση των αρχών για την προστασία της φύσης. Και υπήρχε και εκεί ένας άλλος τόμος τεχνικών πληροφοριών. Γιατί όλα αυτά διότι ακριβώς η, η αυτού του έργου επέβαλε να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή. Οπότε και είχαμε ένα σώρο υπηρεσίες όλα τα κρατημέλη που συμμετέσχουν. Άλλο παραδείγμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Το να μπει κάπου ο σωλήνας που δεν θα κινδύνευε, δεν θα υπήρχε περίπτωση έκρηξης. Και είχαμε τελικά κάποιε εκρήξει που έγιναν ελεγχόμενε από το πολεμικό ναυτικό Φινλανδίας και Σουηδίας. Μα πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εντοπίσει το πού στο βυθό ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει ένα μέρος επικίνδυνο εκεί δηλαδή που δεν θα έπρεπε να πάει ο αγωγός ούτως ώστε να αποφευθεί τυχόν έκρηξη. Τέλος πάντων, ναρκαλίευση και τέ, τέτοιου είδους ε, αλίευση των, των, των, των, παλαιών εκρηκτικών που, που υπήρχαν εκεί, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται τακτικά και θέλω να σας πω επομένως ότι έχουμε εδώ αυτούς οι οποίοι παραπονιούνται για το Nord Stream, όμως εδώ είναι εγγενείς αυτοί οι έλεγχοι αυτέ τις διαδικασίες, όπως σας είπα. Υπάρχει αυτή η διαδικασία και τα κρατή μέλη, τα οποία είναι αρμόδια, ε, δίνουν την άδεια, αλλά, αλλά υπό τον όρο, υπό τους όρους που, που, που τάσουν στον ανάδοχο. Και πολλές φορές πρόκειται και για κάποιες επιπλέον μελέτες τις οποίες ζητούν οι αρχές για να δώσουν την άδεια και θα πρέπει ο ανάδοχος να τις κάνει και σε αυτή την περίπτωση, όπως σας είπα, έχουμε την γερμανική έγκριξη μετά την οποία πρόκυψε ένα θέμα που αφορούσε το κατά πόσο θα υπήρχε προσβασιμότητα σκαφών σε δύο πολωνικά λιμάνια. Γιατί οι πολωνικές αρχές μετά από αυτές τις μελέτες απεφάσισαν ότι στο μέλλον ίσως θα πρέπει να βαθύνουν περισσότερο αυτούς τους λιμένες. Πρόκειται για το Στσέτσιν και το Σίνοβιτ στην Πολωνία. Κατόπιν αυτών Επομένως, αφού δόθηκε η έγκριση για, το, για τον Nord Stream, οι γερμανικές αρχές ανεκάλασαν την έγκριση και θα πρέπει να γίνει καινούργια ανάλυση του κινδύνου. Και, επομένως, η εταιρεία Nord Stream θα έπρεπε να μετακινήσει κατά 12 χιλιόμετρα τον αγωγό. Και σε, άλλο, σε άλλη τοποθεσία θα έπρεπε να βάλει τον αγωγό 1,5 μέτρο πιο βαθιά από όσο στην αρχή προβληθεί. Επομένως, για να απαντήσω στην αξιότιμη βουλευτή, Έχω να πω το εξή. Ναι, επί τη βάση όλων των στοιχείων που επίσημα είχαμε, επί τη βάση του ελέγχου και της εποπτείας που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, ναι, ναι. Θεωρούμε ότι πρόκειται για υποδειγματική διαδικασία και για τη δημοσιοδιαβούλευση και για τα αποτελέσματα τα οποία ε, προέκυψαν και επομένως πρόκειται για ένα έργο και ένα πρόγραμμα το οποίο ε, εξελίσσει την αντίληψη που έχουμε, το, το, την κουλτούρα που έχουμε για τα διασυνοριακά έργα. Αυτά τα είπα και στο παρελθόν. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ότι έγινε συζήτηση μακρά. Κρατή μέλιο, ανάδοχο, όλοι, όλοι μαζί συμμετέχουν και όλοι τους, όλοι τους ανέφεραν ποια είναι η εμπειρία του. Οπότε Όπω ξέρετε τώρα βρίσκεται σχεδόν στη μέση διαδρομή σε αυτό το έργο και επομένω έχουμε 600 χιλιόμετρα αυτού του αγού και χωρίς να έχουν προκύψει τίποτα προβλήματα όσον αφορά παλιά εκρηκτικά, ε, ούτε προβλήματα από τη φύση. Από τον Απρίλιο και μετά που ξεκίνησαν, ε, ξεκίνησε η εκτέλεση του έργου επομένω. Ναι, έγινε δημοσία ακρόαση και επί τη βάση των αναφορών που έχουμε θεωρήσαμε ότι καλά τα πήγαμε, προχωράμε και αντιλούμε συμπεράσματα. Από αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, η οποία παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι ικανοποιεί τους α, ε, ακροατές. Ε, παραμένουν τα ερωτήματα. Α, ε, ξεκινάει τώρα η συζήτηση ο κ. Μαλέζε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απάντησή του στα όσα είπε η κυρία Γέριγκερ. Νομίζω ότι αυτή άλλα σας ρώτησε και εσείς άλλα απαντήσατε. Τα περιβαλλοντικά θέματα του αγωγού αυτού είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι αυτά τα μόνα προβλήματα για τους ανθρώπους της περιοχής. Πρόσφατα ακούσαμε κάποια άλλα ανησυχητικά πράγματα, κάτι που αναφέρατε πολύ σύντομα Κάτι που παραβιάζει την βασική αρχή των ελεύθερων αγαθών και υπηρεσιών, που είναι μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ω το εκτελεστικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόσει τις συστάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα Nord Stream ε, σέβεται το διεθνέ δίκαιο και την αρχή τη ισορροπημένη ανάπτυξη τη Βαλτική θάλασσα. Αυτό σημαίνει ελεύθερη πρόσβαση στα λιμάνια της Πολωνίας. Αυτό αναφέρθηκε πρόσφατα στα ΜΜΕ. Και οι πολωνικές αρχές, από ό,τι φαίνεται, αγνοούν το βάθος στο οποίο βρίσκεται ο αγωγός ε, σε περιοχές από τις οποίες ε, περνάνε αυτά τα πλοία. Είχαμε πει, δηλαδή, αρχικά ότι δεν θα πρέπει ο αγωγός να ενοχλεί τις οδούς των πλοίων. Και παρά τις διαβεβαιώσεις που μας είχαν δώσει, ένας από τους αγωγούς που διασχίζει τη βόρεια, το βόρειο άξονα αυτόν βρίσκεται στα 17,5 μέτρα ε, και παρεμποδίζει έτσι πλοία τα οποία έχουν βήθηση πάνω από 13 ε, μέτρα. 30, συγγνώμη, πάνω από 30 μέτρα. Επομένως αυτό σημαίνει ότι αυτά τα λιμάνια δεν μπορούν να δεχτούν μεγαλύτερα πλοία στο μέλλον και τους παρεμποδίζει την πρόσβαση. Επομένως τα σχέδια που ετοιμάστηκαν ε, πέρυσι δεν είναι σωστά και δεν μπορούμε να δεχτούμε τους ισχυρισμού της Nord Stream. Αυτό θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των λιμανιών στο μέλλον σε σχέση με το λιμάνι Ροστόκ, το οποίο μπορεί να δεχτεί τα μεγαλύτερα πλοία. Το έχουμε θέσει αυτό το θέμα τον Ιούλιο στην Επιτροπή Αναφορών, αλλά το πρόβλημα παρέμενε ανεπίλητο και νομίζω ότι και σήμερα παραμένει ανεπίλητο. Τα ΜΜΕ στις 10 Ιανουαρίου του 2011 ανέφεραν ότι η Nord Stream και οι λιμενικές αρχές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να τοποθετήσουν τον αγωγό βαθύτερα στα σημεία από τα οποία περνάνε τα πλοία. Εγώ φοβάμαι, και δεν είμαι ο μόνος, ότι είναι μια προσπάθεια αυτή για να παρακαμφθεί το πρόβλημα στην πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Επομένως, έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει μια διαδικασία για περιορισμό ε, λόγω του περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών. Να μην, ε, να ξεχνάτε ότι το πρόβλημα της ε, προβληματικής πρόσβασης στα λιμάνια αφορά χωρικά ύδατα μιας χώρας και όχι ε, διεθνή ύδατα και επομένως η Κομισιόν μπορεί να παίξει εκεί κάποιο ρόλο. Θα ήθελα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναφερθεί στο πρόβλημα που ανέφερα και να μου πει αν έχει γίνει μια νομική ανάλυση. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ε, το οποίο ανέφερε η κυρία Γκέριγκερ. Δεν θα το πω διαμακρών, αλλά θέλω να αναφερθώ σε αυτό έτσι δεν τάχει. Την αποζημίωση προς τους αλείς. Θα ήταν άδικο οι Πολωνοί ψαράδες να πληρώσουν τα σπασμένα και να λάβουν 10 φορές λιγότερο από τους ψαράδες, ας πούμε, της Γερμανίας ή της Δανίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μποστινάρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα τετελεσμένο γεγονός κατά κάποιον τρόπον χρησιμοποιώντας τη γαλλική έκφραση φέτα κομπλή διότι η της δανιας ευχαριστω ο κυριος μποστιναρο ευχαριστω κυρια προεδρε ειναι ενα τελεσμενο γεγονος κατα καποιον τροπο χρησιμοποιωντας τη γαλλικη εκφραση φετα κομπλη διοτι η επιτροπη μας λέγει ότι το μισό πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί η εφαρμογή βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής και τι να κάνουμε. Έρχομαι όμως στην έκθεση Μπίσκι και στο περιεχόμενο της, όπου ε, υπήρχαν ε, πολλά ερωτηματικά που δεν έχουν απαντηθεί μέχρι στιγμή. Ε, και καταρχήν όσον αφορά την ε, αξιοπιστία ε, της, ε, της μελέτης. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία έχει αντικρουόμενα συμφέροντα, καλό είναι να το καταγγέλουμε, αλλά κανείς επενδυτής δεν είναι τόσο αφελής, ώστε να να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία η οποία θα αντιτίθεται στα συμφέροντά του. Επίσης δεν έχουμε καμία εγγύηση σε περίπτωση καταστροφής μετά από την ε, καταστροφή που είδαμε με την BP στον κόλπο του Μεξικού. Βέβαια ε, ε, η Nord Stream μας έχει εξασφαλίσει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες και άλλωστε δεν είναι εύκολο να υπάρξει τέτοια εκτάσεως δεύτερη καταστροφή. Αλλά αν οι Αμερικανοί ακόμη ε, τσακώνονται με την BP για ένα διακύδευμα πέραν των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πώς πιστεύουμε ότι κάποιος θα έχει την ισχύ να ζητήσει ε, να αποζημιωθεί σε περίπτωση που επαναληφθεί μια τέτοια δραματική, ένα τέτοιο δραματικό περιστατικό. Ε, ούτε λοιπόν από πρακτικής απόψεως ούτε από θεσμικής απόψεως δεν είναι ασφαλές. Επίσης από πλευράς ασφαλείας ε, διότι υπάρχει το μη συμβατικό στέλεχος της ε, ασφαλείας στη θάλασσα παραδείγματο χάρη όπου έχουμε διάφορα συστήματα που εφαρμόζονται σχετικά με το δίκαιο της θαλάσσης αν ε, εφαρμοστεί ο αγωγός Nord Stream δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Επίσης στη Μαύρη Θάλασσα θα ε, υπάρξει ε, σύντομα μη παρεμφερής εφαρμογή αν δεν διδαχτούμε από το πρώτο εγχείρημα στην Βαλτική. Όσο δε αναφορά τη θέση του Επιτρόπου Ενεργείας έχουμε πλήρη σιωπή. Επίσης η, η ε, Ρωσία δεν έχει ακόμη κυρώσει την συνθήκη ΕΣΠΟ η οποία υποχρεώνει ε, τη χώρα να επιλύσει τα προβλήματα ε, περιβάλλοντος στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λοιπόν, στο δικό μας δηλαδή επίπεδο. Θα ζητούσα από την Επιτροπή να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το θέμα αυτό εις τις συζητήσεις ε, με τη Ρωσία και μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει απάντηση και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο όσον αφορά ε, τον αγώνα μας με τις πολιεθνικές ότι ε, ακόμη είμαστε σε μειονεκτική θέση και πώς θα προχωρήσουμε έτσι. Κύριε Σεμάνσκι, σας παρακαλώ να είσαστε όλοι πιο σύντομοι, γιατί έχω 7 ανθρώπους που θέλουν να απαντήσουν και μετά πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα πρέπει να είμαστε πιο λακωνικοί, αναγκαστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ε, ε, το ψήφισμα του 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται και σε άλλα σημεία όπως τα περιβαλλοντολογικά στο σημείο 15 όπου ζητούσαμε από την Επιτροπή να μας πει ε, αν η επένδυση αυτή θα ήταν συνεκτική με τις διεθνείς συνθήκες και τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ήθελα επίσης να ξέρω ε, αν το πρόγραμμα Nord Stream θα είναι προσβάσιμο εις ε, τις ε, ξένες εταιρείες. Η Gazprom δεν συμπαθεί το κριτήριο αυτό, προσπαθεί να το παρακάμψει και εγώ θα ήθελα να ξέρω εφόσον μιλάμε για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτή αυτής της επενδύσεως, τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγξει τις οικονομικές επιπτώσεις. Επίσης θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται όσον αφορά την, ε, τις επιπτώσεις στην αγορά του φυσικού αερίου. Ζητώ δηλαδή δύο διευκρινήσεις, διότι δεν ισχύει ότι έχει κλείσει η πρόσβαση εις ε, το λιμάνι του Στετίν. Υπάρχει ακόμη η πρόταση αυτή, ε, υπάρχει διαδικασία ε, να παρακάμψει κανείς και να πλεύσει εις το Αμβούργο και ακόμη δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι τα πλοία που θα έχουν βύθισμα 150 μέτρα δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο λιμάνι αυτό. Επίσης Επίσης το άλλο σημείο το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο αγωγός δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο θα οδηγήσει σε μια διαφοροποίηση της αγοράς φυσικού αερίου. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε τις πηγές του αερίου και ε, αυτός ο αγωγός θα οδηγήσει σε ένα μονοπόλιο της αγοράς φυσικού αερίου και θα εξαρτώμεθε όλοι από το ρωσικό αέριο. Εδώ λοιπόν η προσέγγιση της ευρωπαϊκής αγοράς δεν είναι πολύ συνεκτική και δεν έχει καταλάβει η Επιτροπή τη φιλοσοφία ή δεν θέλει να καταλάβει την φιλοσοφία διότι από τις προκαταρκτικές πληροφορίες πληροφορίες που μας έδωσε πρέπει να πω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραβλέπει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να εστιαστεί σε άλλα θέματα και όχι μόνο στα περιβαλλοντολογικά. Κολάς Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες που, από τις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα για το περιβάλλον. Υπάρχουν διαφορετικές αναλύσεις. Υπάρχουν εκείνοι που, όπως είπε η κυρία Γκέργκερ, ε, μιλούν για τις απειλές στο περιβάλλον. Υπάρχουν και άλλες αναφορές που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου εκεί βλέπετε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Επομένως, το θέμα είναι τι να κάνουμε τώρα. Ποια ανάλυση θα θεωρήσουμε ότι είναι πιο αξιόπιστη. Ποιες λαμβάνουν, ποια ανάλυση λαμβάνουμε υπόψη. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό, γιατί στο έργο της Επιτροπής μας ε, αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα πολύ συχνά. Το ερώτημά μου λοιπόν προς την Επιτροπή είναι το εξή. Εσείς, όπως παρακολουθείτε την κατάσταση, αν ε, αποδειχθεί ότι τελικά υπάρχει απειλή και υπάρχει καταστροφή του περιβάλλοντος, θα αποφασίσετε να κλείσετε αυτό το πρόγραμμα, να κλείσετε αυτό το έργο. Μπορείτε να μας πείτε και να δεσμευτείτε σήμερα, ναι, ότι δεσμευόμαστε, ότι αν αντιληφθούμε κάτι τέτοιο, πάρα αυτά θα κλείσουμε, ε, θα σταματήσουμε αυτό το πρόγραμμα και θα κλείσουμε αυτό το έργο. Φυσικά, όπως υπόθηκε νωρίτερα, μπορεί να υπάρχουν, να υπάρχουν κάποιες, κάποιοι κρίκοι της αλήθειας που δεν λειτουργούν, κάποια προβλήματα. Ο ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ένα ολόκληρο πλέγμα ε, υποδομών. Και το Nord Stream αντιμετωπίζεται ως πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Και το νέο πακέτο υποδομών θα το διαπραγματευτούμε ξανά φέτος. Και δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξαναθεωρηθεί ευρωπαϊκό. Αντίθετα, θα προσπαθήσουμε να μην το καταστήσουμε αυτό το πακέτο ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Γιατί? Γιατί. Διάφορες ευρωπαϊκές αρχές και κάποιες ευρωπαϊκές διαδικασίες δεν ακολουθούνται. Στο πακέτο για το μέλλον της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη 2020-2025 αναφέρουμε ξεκάθαρα ότι ζητάμε απόλυτη διαφάνεια για την διακυβερνητική συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία για το Nord Stream και σε θέματα που αφορά τις πιθανές καταστροφές είναι αμφισβητήσιμη, αντίθετη με τις αποφάσεις που πήραμε ας πούμε, για το πρόγραμμα Ναμπούκο. Νομίζω λοιπόν ότι από την αρχή υπήρχαν πολυάριθμες αμφιβολίες για το σχέδιο αυτό, για το έργο αυτό και λαθασμένα θεωρούν ότι ορισμένοι ότι το πρόβλημα είναι της Πολωνίας και της Γερμανίας. Φυσικά υπάρχει το θέμα της γειτονίας και φυσικά το πρόγραμμα έρχεται σε αντίθεση με τα πολωνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά το θέμα τη ελεύθερη πρόσβαση στα ύδατά μα. Αλλά καταρχά και πάνω απ' όλα είναι ευρωπαϊκό αυτό το πρόγραμμα. Και είναι σημαντικό για την εσωτερική αυτή ευρωπαϊκή θάλασσα και για το παράδειγμα που θα δοθεί για άλλα περιβαλλοντικά προγράμματα. Επομένως, θα ήθελα σας παρακαλώ να μου απαντήσετε για το κατά πόσο θα κλείσετε αυτό το έργο, θα σταματήσετε αυτό το έργο, αν χρειαστεί, και να μου απαντήσετε και σε ερωτήματα που αφορούν κυρίως τον Επίτροπο Ενέργειας. Ο Επίτροπος θα ζητήσει κάποια αλλαγή των συμβολέων, των συμβάσεων, σε περίπτωση που υπάρξουν αυτά τα προβλήματα τα οποία σας αναφέραμε. Θα μιλήσω λετωνικά. Λοιπόν, ας επωφεληθώ από την ε, διερμηνία που έχω σήμερα, ας μιλήσω τη γλώσσα μου. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να εξετάσουμε αυτό το θέμα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Από περιβαλλοντική σκοπιά. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Υπάρχουν κάποια πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που υπάρχουν ακόμα στις θάλασσες, στη θάλασσα αυτή, εν περιπτώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει μια τρομακτική απειλή λόγω αυτών των παλιών πυρομαχικών στη Βαλτική. Έχουν γίνει μοιραία ατυχήματα. Σε, θυμάστε περιπτώσεις, ίσως να γνωρίζετε περιπτώσεις όπου ε, ψαράδες έχουν ψαρέψει παλιά τέτοια πυρομαχικά και έχουν εκραγεί αυτά. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ε, έγινε η πρόταση για το Nord Stream, θεωρήθηκε ότι οι εταιρείε που θα έχουν μετοχέ σε αυτό το πρόγραμμα Nord Stream θα επιλύσουν να θα προσπαθήσουν και θα συνεισφέρουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Θεωρούσαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους τους για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτό που ακούμε όμως σήμερα και, ότι και αυτά που διαβάζουμε στον τύπο δείχνουν ότι η οδή, η οδός μάλλον που επιλέγει, καθαρίστηκε και όλα είναι μια χαρά. Αλλά όμως το πρόβλημα δεν έχει ξεπεραστεί, γιατί υπάρχουν και άλλες περιοχές στη Βαλτική, που ψαρεύουν οι ψαράδες και εκεί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα, ε, επειδή εστιάσαμε την προσοχή μας μόνο στον δρόμο από τον οποίο περνάει ο αγωγός, τι γίνεται με την υπόλοιπη Βαλτική η Κομισιόν θα πρέπει να δει αυτό το θέμα έτσι με, μια πιο ανοιχτή, πιο πλατιά ματιά. Γιατί όλα αυτά τα θέματα συνδέονται με το έργο του Nord Stream. Και στην έκθεσή μας και στο ψήφισμά μας θα πρέπει να αναφέρουμε το θέμα των παλιών πυρομαχικών, των παλιών όλμων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Κάποια στιγμή πρέπει να το επιλύσει αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άπαξ και διαπαντό. Κάνω έκκληση λοιπόν στον εισηγητή μα να αναφερθεί, να αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα που, για τα οποία μίλησα και να τα συμπεριλάβει στην έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Βαλτική είναι ε, μία από τις ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές που είναι πολύ ευαίσθητη στη ρήπανση, πολύ περισσότερο από ότι η ε, Μεσόγειος και ο κύριος Μποστινάρο ανέφερε τι έγινε στον κόλπο του Μεξικού. Αλλά όσον αφορά τη Βαλτική είναι μία περιοχή πάρα πολύ ευαίσθητη και πιστεύω ότι αυτό έπρεπε επίσης να ληφθεί υπόψη διότι κοιτούμε μία περιοχή θαλάσσια η οποία πεθαίνει εάν κάτι δεν γίνει ή εάν υπάρξει ρήπανση. Οπότε θα έπρεπε να κοιτάξουμε την ιδιάζουσα κατάσταση της βαλτικής περιοχής. Ο κύριος Γιάρ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα έχω τέσσερα ερωτήματα συμπληρωματικά. Ε, καταρχήν, σε τέτοιες ε, μεγάλες, ε, μεγαλεπίβολες καταστάσεις πρέπει να υπάρχει μία μελέτη σκοπιμότητος και πρέπει είτε να θεωρήσει κανείς ότι θα αποτύχει το πρόγραμμα ή είναι ανεκτές και μπορούν να αντισταθμιστούν οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Θα, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή ποιος θα καταρτήσει αυτή τη μελέτη για να είναι κάποιος ανεξάρτητος και να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Μετά, όσον αφορά το σενάριο καταστροφής, δεν φτάνει να μου λέει κάπως ότι έχουμε αρκετά χρήματα να διαθέσουμε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια τέτοια καταστροφή γιατί είδαμε από την ε, ε, καταστροφή του Μεξικού ότι οι μηχανικοί δεν είχαν προβλέψει νέες καταστάσεις και δεν είχαν τα ενδεδειγμένα τεχνικά μέσα για να παλέψουν. Οπότε ε, έχουμε στη μελέτη αυτή λάβει επίσης και το worst case σενάριο δηλαδή την περίπτωση μιας καταστροφής. Επίσης κάτι άλλο που ελέγχει είναι πολύ σημαντικό. Μέσω αυτού του αγωγού πρόκειται πρόκειται να κινδυνεύσουν τα λιμάνια της Βορείου Θαλάσσης όσον αφορά το βήθισμα των πλοίων, δηλαδή μπορεί αυτό να επηρεάσει τη βιωσιμότητα λιμανιών της Βορείου Θαλάσσης και επίσης ε, όσον αφορά την, ε, ε, την κατάσταση των αλλιέων υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις στην περιοχή εκεί κυρία Γκέριγκε τα τελευταία Ευχαριστώ Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ήταν εκτός θέματος Άλλες ερωτήσεις έκανα εγώ, σε άλλες απάντησε η Επιτροπή. Ας περιμένουμε την ε, επόμενη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω να είναι εντός θέματος και πιο λεπτομερής. Έχω άλλη μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει ξανά και ξανά ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν νομικά μέσα, ένδικα μέσα, για να ζητήσουμε ανεξάρτητη αξιολόγηση, ανεξάρτητη μελέτη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι αυτή η μελέτη που έκανε ο επενδυτής είναι τέλεια. Εγώ θα έλεγα να τροποποιήσει τη σχετική οδηγία του 1985 παρά να μας επαναλαμβάνει αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι μια καινοτομία. Είναι το πρώτο στο είδο του. Κανένας δεν έχει ξαναφτιάξει τέτοιου είδου αγωγό ε, στο βυθό της θάλασσας, ε, που είναι μια πολύ ρηχή θάλασσα. όπου δεν κυκλοφορούν αρκετά τα νερά. Τα νερά είναι ήσυχα, δεν υπάρχει μεγάλη ροή και αν γινόταν κάποιο ατύχημα θα είχε δραματικές και καταστροφικές επιπτώσεις. Άρα θα πρέπει να βρούμε τα νομικά εργαλεία. Δεν ξέρω. Αν την πρόσφατη έκθεση του 2010 της Nord Stream για το monitoring, η οποία ετοιμάστηκε ε, ενώ το πρόγραμμα ήταν στο μέσο της ζωής του. Στην έκθεση αυτή λέγεται ότι η Nord Stream θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το οικοσύστημα της ε, Βαλτικής θάλασσας αρκετές εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του αγωγού και μερικές μέρες, μερικές φορές, ε, μέρες μετά την ολοκλήρωση της οικοδόμησης, λέει, του αγωγού. Τι συμπεριφορά είναι αυτή, μερικές μέρες θα την παρακολουθεί ή μερικές εβδομάδες, τι είναι αυτό το πράγμα δεν συμφωνούμε με αυτή την έκθεση. Είναι επαγγελματική δηλαδή αυτή η έκθεση που ετοίμασε τώρα η Nord Stream. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής και του ζητάω για λόγους περιορισμού χρόνου να απαντήσει με τρόπο λακωνικό. Την πιο λεπτομερή απάντηση θα ήθελα να μας τη δώσει γραπτός. Το λέω σε όλους. Έχουμε μία ώρα καθυστέρηση σε σχέση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν θέλουμε να προωθήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών, θα πρέπει να περιορίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και, και τα δικό μας, ας πούμε, τη δική μας όρεξη για μονοπόληση του μικροφώνου. Λίγα λεπτά για την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνω την περιπλοκότητα του προβλήματος, γιατί και για μας ήταν ένα τεράστιο πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ήταν το πρώτο στο είδος του, αλλά καταλάβετε με, όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα, ε, όλοι προσεγγίζουμε με τον τρόπο τα θεσμικά θέματα. Ε, η Σύμβαση ΕΣΠΟ και το Δίκαιο για τα Περιβαλλοντικά Θέματα προβλέπει μια διαδικασία που είναι υπό την αιγίδα των κρατών μελών για πολύ καλούς λόγους, για πολύ ευνόητους λόγους. Ακούσατε όλα αυτά τα θέματα. Είναι αδύνατον οποιοδήποτε σώμα, οποιοδήποτε φορέας να εντοπίσει όλα αυτά τα θέματα που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Κομισιόν δεν μπορεί να πάει στους Φιλανδούς και να τους πει «Όχι, έτσι θα πρέπει να, να να εκραγούν ελεγχόμενα τα, τα πυρομαχικά ή ξέρω εγώ έτσι να προστατεύσετε τη φύση». Ας σας μιλήσω για αυτή τη διαδικασία πολύ σύντομα. Η οδηγία λέει ότι όταν ένας ανάδοχος ζητάει να υπάρξει μια άδεια για ένα πρόγραμμα και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε έναν ιδιωτικό, ένα ιδιωτικό πρόγραμμα που αφορά τα κράτη-μέλη όπου θα λάβει χώρα το πρόγραμμα αυτό στην ε, αποκλειστική οικονομική του ζώνη και στα χωρικά του ε, ε, ύδατα και ζητάνε άδεια αυτέ οι εταιρείε, αυτά τα κράτη-μέλη για να δώσουν την ε, άδεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το νομικό εργαλείο στο οποίο όλοι αναφερόμαστε. Αυτή τη μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωση υπό την αιγίδα μας, κάτι που είπα και στην ε, απάντησή μου, και να ε, χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν και την σύμβαση ΕΣΠΟ. Ε, δηλαδή, ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να δώσει τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχέ που αυτές του ζητάνε για να αξιολογήσει για να αξιολογηθεί το, ε, το πρόγραμμα. Και με βάση το άρθρο 5 της οδηγίας, ο ανάδοχος θα δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες. Ποιος δίνει λοιπόν τις πληροφορίες είναι σαφές. Ο ανάδοχος. Κανένας ανεξάρτητος φορέας που ήταν δύσκολο να θεσπιστεί και να δημιουργηθεί και το εξηγώ γιατί. Γιατί ο ανάδοχος δίνει τις πληροφορίες. Αλλά αυτές οι πληροφορίες εξετάζονται. Και είναι δύσκολο να πούμε ότι η πληροφορία τελικά δεν είναι αξιόπιστη, γιατί εξετάζεται αυτή η πληροφορία. Γιατί οι περιβαλλοντικές αρχές εξετάνε τα τεχνικά θέματα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις επίσης και το κοινό εξετάζει επίσης όλες αυτές τις πληροφορίες. Η οδηγία τι λέει εν συνεχεία. Λέει ότι η αρχή υπεύθυνη για την άδεια του έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες αυτές τις πληροφορίες και να λάβει την ε, κατάλληλη απόφαση. Και όπως είπε κάποιος βουλευτής, δεν, δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή η περιβαλλοντική μελέτη είναι αρνητική δεν την κάνω, τα κράτη-μέλη ούτως ή άλλως μπορούν να δώσουν την άδεια και να την συναρτήσουν από τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Και σας διαβεβαιώ ότι όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν αυτή τη διαδραστική διαδικασία με την Nord Stream. Κάθε τόσο καλούσαν την Nord Stream να τους δώσει περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες στις τεχνικές, αρμόδιες τεχνικές τους αρχές. Δόθηκαν άπειρες πληροφορίες. Ανταλλάγησαν ε, τέτοια στοιχεία μεταξύ της Nord Stream και των αρμοδίων τεχνικών αρχών των κρατών μελών. Στη Γερμανία μάλιστα είχαμε δύο δημόσιες αρχές που έπρεπε να δώσουν άδεια και έγκριση. Αυτά με την νομική διαδικασία. Είμαστε σε φάση αναθεώρηση της οδηγίας για την ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα έρθει σε εσά το σχετικό κείμενο και θα έχετε την ευκαιρία να πείτε ότι δεν θα πρέπει ο ανάδοχος Φερρυπή να δίνει τις πληροφορίες, αλλά ένας ανεξάρτητος φορέας. θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Τώρα για τα υπόλοιπα θέματα, σύντομα. Το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα στις πρώτες φάσεις του, εκεί δηλαδή μέχρι να οικοδομηθεί ο αγωγός. Αυτή τη στιγμή δημιουργηθεί ο αγωγός, υπάρξει και μπει ο αγωγός, δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Τώρα, οι αποζημιώσεις των αλλιέων προβλέφθηκαν ούτω ώστε να τους αποζημιώσουμε για την περίοδο της προετοιμασίας που δεν μπορούν να ψαρεύουν, κατά την οποία δεν θα μπορούν να ψαρεύουν. Οι αποζημιώσει επίση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Κομισιόν, και δεν έχω την απάντηση, θα προσπαθήσω να τη βρω, αλλά δεν μπορεί η Κομισιόν να καθορίσει τις αποζημιώσεις προς τους αλείς. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν. Τώρα για τα λιμάνια, τα οποία αναφέρατε πολλοί από εσά. Σας εξήγησα ότι όταν δοθούν οι άδειε, οι πολωνικές αρχές ε, υπέβαλαν σχέδια για να αυξηθεί το βάθος του λιμανιού. Και μόνο σε αυτή τη φάση οι αρχές ξανά είδαν το θέμα και αυτό που είπατε είναι σωστό. Ότι ο Nord Stream μαζί με τις λιμενικές αρχές της Γερμανίας και της Πολωνίας θα δημιουργήσουν μια ομάδα εργασία που θα αρχίσει να εργάζεται το Φεβρουάριο, τόσο ώστε να βρεθεί ένα θέμα, ε, μια λύση για το θέμα του βάθου του λιμανιού. Το θέμα αυτό λοιπόν το εξετάζουν οι αρμόδιοι, Πολωνοί και Γερμανοί. Ε, για τα υπόλοιπα μπορείτε να βρείτε απαντήσεις ε, στην ανακοίνωση Μην ξεχνάτε λοιπόν ε, ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα που είναι σε φάση προετοιμασίας, ε, όπως το Ναμπούκο κτλ. Ε, είναι αδύνατο για κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα να κάνουμε την ίδια προσπάθεια, να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με αυτή του Nord Stream. Σας ευχαριστώ. Το θέμα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, εξού και πολλές ερωτήσεις. Σας λέω εκ των προτέρων ότι σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις των συντονιστών θα θέσω το θέμα της στάσης που πρέπει να έχει η Επιτροπή μας όταν αντιμετωπίζουμε, ε, όπως αυτή την περίπτωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, θέματα τα οποία θέτουμε και στα οποία δεν συνέχεια. Το πρόβλημα δεν είναι η σύγκρουση μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ε, στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που εμφανίζεται ξανά και ξανά. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο για να σεβαστούμε, όπως σας είπα προηγουμένως, τους πολίτες. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές, θα πρέπει να τις... και προσπαθούμε όλες αυτές τις πολλές αναφορές να τις... Θα πρέπει τώρα, λόγω του ότι καθυστερήσαμε, να τις εξαντλήσουμε στο μισόχρονο από ό,τι είχαμε προβλέψει. Σας παρακαλώ, τώρα, για τις επόμενες αναφορές, τρία λεφτά για τους πολίτες, ε, ένα λεπτό για τους βουλευτές, όχι παραπάνω, γιατί αλλιώς θα διεκπαιρέσουμε όλες τις αναφορές. Και περνάω στην αναφορά 16 και δίνω το λόγο στην Ιρένα Ρογκόσκα. Όχι, εξ ονόματός της μιλάει ε, η κυρία Βασνιέσκη, για τρία λεφτά όπως σας είπα. Ε, ευχαριστώ. Είμαι η κυρία Ρογκόφσκα, ε, που κατήρτισε την ε, αναφορά 46 εκπροσωπώ την ε, περιοχή μου σαν ε, επικεφαλής της κινήσεως για να σταματήσουμε την, το υπαίθριο λιγνητορυχείο οτι ε, ε, αντιλαμβάνομαι ότι προβλέπεται η δημιουργία ενός λιγνητορυχείου επιφανίας. Πριν 18 χρόνια ξεκίνησε ε, η κατασκευή αυτή για την εξόριξη λιγνίτη με την προστασία της σοβιετικής, ε, ε, του σοβιετικού στρατού και δεν υπήρχε τότε ε, αυτοδιάθεση αλλά τώρα είμαστε στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα μεγάλο εγχείρημα όπου και οι μικρές κοινότητες μπορούν να προασπίσουν τα δικαιώματά τους. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και ε, από το 2007 είδαμε ότι ε, προβλέπεται να ξαναξεκινήσει η εξόριξη ε, λιγνίτη στην περιοχή αυτή παρόλο που αντιτίθενται από το 78 δεκάδες χιλιάδες ατόμων τότε ο πληθυσμός της περιοχής έχει αυξηθεί έχει έχει δημιουργηθεί μία υποδομή και χρησιμοποιούμε τους δικούς μας πόρους αλλά και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η εφαρμογή των προγραμμάτων για την εξόριξη του λιγνίτη σημαίνει ότι θα υπάρξει η ε, δημιουργία του μεγαλύτερου ορυχείου επιφανείας ε, στην Ευρώπη και ε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στους πολίτες αν θα είναι ασφαλής διότι ε, δεν έχουμε απάντηση στις αιτήσει που έχουμε απευθύνει στην ε, πολωνική κυβέρνηση. Γι' αυτό και έγινε ένα δημοψήφισμα το 2009. Το δημοψήφισμα ήταν ε, έγκυρο και δεσμευτικό, δεν ξέρουμε όμως εάν θα εφαρμοστούν τα απορίσματα και ε, η νομοθετική εργασία δείχνει ότι υπάρχει ακόμη απειλή του λιγνητορυχείου επιφανείας και ε, το 95% των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα ήταν υπέρ αυτής της δημιουργίας. Κοιτάξτε, υπάρχει και άλλη παρέμβαση, πρέπει να συντομεύετε. Θέλω λοιπόν ε, να προασπίσουμε τα, τα ε, δικαιώματά μας ε, και απευθύναμε ένα αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούμε από την Επιτροπή σας να αναλάβει κατά προτεραιότητα την έρευνα και να προβεί στην αποστολή ενός ενός κλιμακίου έρευνας για να μπορέσει να βοηθήσει τους πελίτες. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο ο επόμενος ομιλητής. this one. E, e, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εν ονόματι μίας ομάδας περιβαλλοντολόγων θα ήθελα να παρουσιάσω την αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών ζημιών που θα δημιουργήσει ε, το λιγνητορυχείο εάν υπάρξει ένα ορυχείο επιφανίας και θέλω να ε, κάνω δύο γενικές ερωτήσεις καταρχήν. Πρώτον ε, ότι θα δημιουργηθεί το ορυχείο αυτό ενώ υπήρχαν άλλες εναλλακτικές λύσεις και δεν έγινε συζήτηση των εναλλακτικών λύσεων. Δεύτερον, παρόλη την ε, ύπαρξη ε, μίας ε, περιοχής επί πολύ καιρό δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση της περιβαλλοντολογικής κατάστασης της περιοχής και πρόκειται να είναι ένα τεράστιο ορυχείο 140 τετραγωνικών χιλιόμετρων το οποίο θα επηρεάσει μία περιοχή 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων όσο αναφορά τις τα υπόγεια ύδατα και θα προκαλέσει μία σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον και σε σημαντικές ε, πρακτικές περιοχές, πέντε περιοχές Natura 2000 που προστατεύονται από την οδηγία για τα οικοσυστήματα θα, θα χρειαστεί κιόλας να διαλυθούν δύο ο, περιοχές με δάση που συνδέονται με τις προστατευόμενες περιοχές ε, θα καταστρέψει ένα δάσος ε, μοναδικό χώρο λιμνών και βεβαίως και ε, πολλά ποτάμια. Βλέπετε εδώ τον διάδρομο που περνά από την Γερμανία προς Ανατολάς και πώς δάση υπάρχουν, πόσες προστατευόμενες περιοχές περιβαλλοντολογικές που διέπονται από την προστατευτική πολωνική νομοθεσία σχετικά με τις επιταγές της Natura 2000. Βλέπετε εδώ τον διάδρομο δασών ο οποίος καταστρέφεται και με πράσινο βλέπετε ε, το χώρο του λιγνητορυχείου και γύρω το χώρο ο οποίος πρόκειται να επηρεαστεί. Εδώ βλέπετε πόσο καταστρέφονται δάση τα οποία βρίσκονται ε, μεταξύ πόλεων ε, που ε, έχουν συνολικά 200.000 κατοίκους και αυτό δείχνει την καταστροφή της περιοχής. Θα υπάρξει και η καταστροφή ε, των ε, ε, χώρων όπου στεγάζονται διάφορα πτηνά θα καταστραφεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας και κατά τη γνώμη μας αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι σύμφωνα με τις προ, ε, τους υπολογισμούς μας το περιβαλλοντολογικό κόστος ενός τεραστίου τέτοιου ορυχείου θα είναι υπερβολικό ε, για να μπορέσει το πρόγραμμα να είναι περιβαλλοντολογικά ασφαλές. Αντιθέτως θα υπάρχει μία σαφής απειλή ε, για πολλά είδη στην ανατολική και δυτική πλευρά και τη η δυνατότητα να αποδημήσουν από Γερμανία προς Ανατολάς τα ε, ίδια αυτά. Θα έπρεπε λοιπόν ε, να υπάρχει μία ε, πολυσχηδής ε, μελέτη καταρχήν για να αξιολογηθεί το, η κατάσταση του περιβάλλοντος και στο μέλλον και μετά να γίνει μία μελλοντική περιβαλλοντολογική μελέτη επιπτώσεων διότι η πρώτη δεν βασίζεται σε πλήρη στοιχεία και αυτό βέβαια μπορεί να ερμηνευθεί ε, ως λόγο για τον οποίο υπήρχε θετική χορήγηση αποφάσεως. Η κυρία Κοφλώσκα τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως και θα μπορούσατε να, συμπεράσετε από αυτά το οποία είπε η υποβαλούσε την αναφορά ότι ε, απευθυνόταν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε ζητηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα. Και για αυτό ε, υπήρξε η ευκαιρία στην προηγούμενη επαφή μας να λάβουμε υπόψη τα όσα είχαν να πούν οι πολωνικές αρχές για το θέμα. Επομένως, ευθύ εξ αρχής σας λέω ότι είχαμε εδώ το, θέμα ήταν ε, αυτές οι εγκαταστάσεις στην Σιλεσία, για τις οποίες ακόμα δεν έχει δοθεί έγκριση. Και από ό,τι γνωρίζουμε, αυτές οι επιφυλάξεις των ε, υποβαλλόντων την αναφορά αναφέρονται στην ε, ενεργειακή στρατηγική της Πολωνίας ε, μέχρι το 2020 όπου Αυτά τα κοιτάσματα λιγνίτη ε, προστατεύονται σε σχέση με έργα επιφανείας που θα ε, γινόντουσαν κοντά στα κοιτάσματα. Οπότε ε, θεωρήθηκε ότι θα υπήρχαν επιπτώσεις σε τοποθεσίες καλυπτόμενες από το Natura. Έχουμε επομένω εδώ πέρα δύο οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που συντρέχουν πρώτα-πρώτα. Έχουμε την ε, περιβαλλοντική αξιολόγηση, την, την οδηγία περιβαλλοντική αξιολόγηση και δεύτερον έχουμε μια άλλη οδηγία όσον αφορά την ε, προστασία πανίδας και χλωρίδας και επίσης συγκεκριμένων προστατευομένων φυσικών χώρων. Έγινε η ανάλυση μέσω των δεδομένων από τις αρχές και σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια τέτοια μελέτη αξιολόγησης η οποία θα έπρεπε επίσης να περάσει και από ε, δημοσία διαβούλευση. Επίσης το σχετικό έγγραφο αυτό δηλαδή που περιέχει την στρατηγική μέχρι το 2030 είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει το πώς θα ασκηθεί η περιβαλλοντική πολιτική. Δεν ασχολείται αυτό το έγγραφο με κάποιο συγκεκριμένο έργο ή πρόγραμμα. Σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο θα πρέπει αυτά τα προγράμματα και έργα να ενταχθούν ε, σε κάποια νομοθετήματα που αφορούν, που αφορούν την ε, περιφερειακή χωροταξία. Όλα αυτά επομένω ε, σχετίζονται με τις οδηγίες που σας προανέφερα. Εμείς αναλύσαμε αυτό το στρατηγικό έγγραφο, κάναμε σύγκριση με τις οδηγίες και είπαμε ότι είναι αβάσιμο τώρα αν θεωρεί κανεί το ότι υπάρχει εδώ παραβίαση διατάξεων της οδηγίας. Έχουμε τώρα το άρθρο 6 το οποίο συντρέχει το και το οποίο ορίζει ότι οποιοδήποτε έργο, όπως το έργο εν προκειμένου, που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε κάποιο χώρο που καλυπτόμουν από το Natura, θα πρέπει για να προχωρήσει ως πρόγραμμα, ως έργο, να υπάρξει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα δε με την πολωνική κυβέρνηση, αυτά τα κοιτάσματα λιγνίτη θα πρέπει να για να, προχωρήσει το έργο τέλο πάντων σε αυτά τα, τα μέρη από του Νατούρα, θα πρέπει να ε, επιτρέπεται αυτό από τα νομοθετήματα που προαναφέραμε. Επομένως θα πρέπει να εξεταστεί αν υπάρχει κάποια περιφερειακή αστονομοθεσία στη χώρα που να επιτρέπει τέτοιου είδους ε, έργα σε σχέση με αυτά τα κοιτάσματα λιγνίτη. πρόεδρο. Συνεχίζουμε η κυρία Ολάσκα. Σας ευχαριστώ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, διότι μιλούμε για κάποια επένδυση, κάποιο έργο που θα ολοκληρωθεί σε 20 χρόνια. Δεν ξέρουμε επομένω τι θα απογίνει. Ε, μιλούμε τώρα για κάποιο, κάποια στρατηγική, για κάποιο προγραμματισμό ε, η δε κυβέρνηση λέει ότι θα αποφασίσει ό,τι χρειάζεται να αποφασιστεί. Επομένως τώρα αναδύεται ένα άλλο θέμα. Το ότι η κυβέρνηση δεν ξέρει καν εάν θα μπορέσει, αν θα έχει τους πόρους να προχωρήσει αυτό το έργο. Ίσως δε, επιπροσθέτως, αλλάξει η όλη σύλληψη για τέτοια έργα. Επομένως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό επομένω. Ε, ότι δηλαδή έτσι μπλοκάρονται έργα και προγράμματα. Αυτό είναι πρόβλημα και είναι ικανός λόγος να υποστηρίξουμε αυτή την αναφορά. Ο επόμενος. Η επομένη μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω, λέει κυρία Γένιγερ, να ερωτήσω την ε, Επιτροπή γιατί αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τα πολωνικά επιχειρήματα. Είναι κατά κάποιο τρόπο διάδικος εδώ. Εμπλέκεται άμεσα η πολωνική κυβέρνηση. Θα πρέπει να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Έχουμε το δημοψήφισμα δεδομένο. 95% σε αυτό το δημοψήφισμα από τους κατοίκους της περιοχής είπαν όχι. Όχι σε αυτή την εγκατάσταση εξόριξης του λιγνίτη. Ήταν πρόβλημα και η τάξη μεγέθους για αυτό το λιγνητορυχείο. Γιγαντιαίο θα ήταν. Γι' αυτό και υπήρχαν αυτοί οι φόβοι και επιφυλάξεις και προβληματισμοί. Συνάδελφοι, αφού 95% του κόσμου είπαν όχι. Όμως χωρίς να έχουν αντίρρηση με την περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη της περιοχής. Γιατί να μην αναζητηθούν εναλλακτικέ λύσεις. Με κατακλείδη κυρία Πρόεδρε, έχω μία ερώτηση επιπλέον. Ξέρω ότι πιέζει και ο χρόνος. Θα ρωτήσω τον κύριο καθηγητή πώς αξιολογεί την μελέτη επιπτώσεων των πολωνικών αρχών. Επίσης και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών θέλω να μου πούν τι προέκυψε όσον αφορά την ε, διαβούλευση που αφορά την ενεργειακή στρατηγική. Ο επόμενος. Εγώ είμαι ευρωβουλευτής και ζω στην εν λόγω περιοχή, λέει ο κύριο Μπόρι. Εδώ πρόκειται για το μεγαλύτερο κοίτασμα λιγνίτη που υπάρχει στον κόσμο. Ε, αν το λιγνητορυχείο προχωρήσει, θα έχουμε ανοίγει στο βλάβη στο περιβάλλον. Θα πρέπει όπως έχει γίνει αλλού και η Πολωνία να περιορίσει τις εκπομπές διοξείδου του άνθρακος. Κατά τη γνώμη μας, δεν έγιναν οι δημόσιες διαβουλεύσεις όπως έπρεπε. Θα πρέπει η διαδικασία να επαναληφθεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν παραδεκτά τα όσα εδώ ισχυρίζονται σε αναφορά. Η δε κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει ευθύ αμέσω στην εκτέλεση του έργου. Θα πρέπει να έχουν περιορισμοί όσον αφορά την εκμετάλλευση αυτού του κοιτάσματο. Επίση, μπλοκάρεται η ανάπτυξη τη περιοχή λόγω του ανθρακοριχείου. Δηλαδή, επηρεάζεται άμεσα η ζωή, το επίπεδο ζωή των ε, κατοικούντων την περιοχή. Άρα, να κάνουμε αποδεκτή αυτή την αναφορά. Να πούμε ότι θα πρέπει η Πολωνία να ξανακάνει ε, ορθά τις ε, διαβουλεύσεις και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι μακρόπνοες επιπτώσεις ε, περιβαλλοντικές και γενικότερα. να... Κάτι γνώμη μου είναι σαφές ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Δεύτερον, ε, ε, ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη την τάξη μεγέθους αυτού του έργου που θα είναι το μεγαλύτερο αυτού του είδους στην Ευρώπη, εγώ θα πρότεινα να στείλουμε ως Επιτροπή Αναφορών επιστολή στην Πολιτική Κυβέρνηση, να μας παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες για τη στρατηγική, για την δυνατότητα υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Εδώ, από αυτό εδώ το ψηφιδωτό, λείπουν πολλά κομματάκια. Επίσης, είναι προφανές ότι για ένα τέτοιο φαρονικό έργο, αν δεν έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, τότε τίθεται κινδύνο και η βιοπικιλότητα και το Natura 2000 και το φυσικό προστατευόμενο περιβάλλον και για αυτό θέλω να απευθυνθώ στους δύο ε, υποβάλλοντες αναφορά να μας πούνε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση αλλά και στο περιβάλλον άκουσα και τον αξιότιμο κύριο καθηγητή και η απάντηση είναι ξεκάθαρη θα είναι τερατώδες οι συνέπειες γιατί μιλούμε εδώ για ένα έργο το οποίο θα γίνει στο μέλλον. Επομένως τώρα φαίνεται πρόημο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε αυτή την επιστολή στην πολωνική κυβέρνηση, να μας παράσχει τις απλές πληροφορίες, η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προσέξει πάρα πολύ τις εξελίξεις που θα σημειωθούν, διότι για ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί κανείς ε, να θεωρήσει ότι αυτό που μετράει είναι τα, τα λεφτά, money talks. Είναι τέτοιον διαστάσεων το έργο που αυτό το επιχείρημα είναι παράδεικτο. Ευχαριστώ κύριε Μποσινάρου για την απάντηση τώρα. Θα δώσουμε για ένα λεπτό το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί να απαντήσει και στι υποβληθείς ερωτήσεις. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα πρώτα τα επιχειρήματα, οι ισχυρισμοί που ακούσαμε αφορά, αφορούν την πολωνική κυβέρνηση και όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί σα βεβαιώνω ότι θα παρακολουθήσουμε την εκτέλεση του έργου και θα επαγρυμνήσουμε για την τήρηση του κοινοτικού δικαίου. Τώρα, όσον αφορά τις επικρίσεις ότι δεν είχαμε σωστές ε, ε διαβουλεύσεις, να σας πω ότι σήμερα τις που έχουμε δεν, δεν υπάρχουν στοιχεία για το ότι είχαμε τέτοιου είδους παραλήψεις από πλευρά πολωνικών αρχών. Και γι' αυτό και πιστεύω την προσοχή στο γεγονό ότι η συντρέχουσα οδηγία επιτάσσει υποχρεωτικά να γίνονται αυτές οι διαδικασίες διαβούλευσης. δε υποχρέωση των πολωνικών αρχών είναι να οργανώνεται η διαβούλευση. Εάν όμως υπάρχουν στοιχεία ότι δεν έγινε σωστή διαβούλευση πρέπει να ξαναγίνει. Και τώρα στον, στον Δήμαρχο ο λόγος, λέει η Πρόεδρος. Εγώ έχω να σας ενημερώσω για το ότι υπήρξαν κάποιοι πόροι που εκταμιέθηκαν για να καλυφθούν 45.000 άνθρωποι και για κατασκευή κάποιων νοσοκομιακών μονάδων. Ακριβώς λόγω του ότι ζούμε εν μέσω κοιτασμάτων λιγνίτη και επίσης και για σχολεία πήραμε κάποια χρήματα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για παιδικούς σταθμούς για την πολιτική καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού για διαγνωστικές δραστηριότητες ιατρικές για την πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου Έχουμε επίσης ε, κάποια άλλα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την εξεργασία των λιμάτων και ενέργειες των εγκαταστάσεων. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τα οποία διατέθηκαν για την ε, κατασκευή υπονόμων και θεωρήθηκε ότι πρώτα πρώτα θα φτιάξουμε αυτό το λιγνωργείο και στη συνέχεια θα έχουμε μετά την ε, κατάργηση αυτού του δικτύου υπονόμων. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα στην εξέταση της αναφοράς και θα πρέπει όσο έχουμε χρόνο να έρθουμε σε επαφή με τις πολωνικές αρχές. Και είπαμε ότι δεν έγιναν σωστά αυτέ οι διαβουλεύσει και μόλι θα πρέπει οι για να μα παράσχουν περισσότερε λεπτομέρειε και στοιχεία. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το στρατηγικό έγγραφο και κατά πόσον είναι βάσιμε οι ανησυχίε που διατυπώθηκαν. Οπότε, παρακαλούμε να συνεργαστεί η Επιτροπή και έτσι να κάνουμε αυτό το οποίο αποφασίζαμε σήμερα. Πάμε τώρα στην αναφορά υπαριθμό 17. quindi do direttamente la parola al rappresentante della Commissione. Eh. Στην αναφορά υπαριθμό 17 μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διαφωτίσει, μια που δεν παρήσατε εδώ ο υποβάλλοντας αναφορά. Θα είμαι σύντομος κύριε Επίτροπε, ιδίως ε, όσον αφορά την ε, αίτησή σας να είμαστε σύντομοι. Εδώ πρόκειται ε, για ε, τον, την περίπτωση ενός Γάλλου υπηκόου ο, ο οποίος αναφέρεται εις ε, την ε, εγκατάσταση ε, επεξεργασίας λιμάτων του Μπεζιέ που κατά τη γνώμη του προκαλούν περισσότερες επιπτώσεις και επιδεινώνουν την κατάσταση. Τρεις εβδομάδες μετά την υποβολή της εκθέσεως ζητήθηκε από την Επιτροπή όχι μόνο να εξεταστεί το θέμα αλλά συγχρόνως να βελτιωθεί η ακατάλληλη μονάδα επεξεργασίας λιμάτων ότι έπρεπε να επεξεργάζονται και τα ακάθαρτα ύδατα που δημιουργούσαν τα προβλήματα. Μία τέτοια τροπολογία έπρεπε ε, να προκαλέσει ε, μία υποχρεωτική ε, εξέταση επιπτώσεων όπου οι πολίτες όπως και ο ετών έπρεπε ε, να ε, πούν τη γνώμη τους σχετικά με ε, το θέμα της επεξεργασίας των αστικών λιμάτων. Οι γαλλικές αρχές λοιπόν έπρεπε να σεβαστούν ακριβώς τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις η Επιτροπή εξέτασε επίσης εάν η ε, αίτηση αυτή, η αναφορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως λύματα που δημιουργήθηκαν από την ακατάλληλη μονάδα επεξεργασίας στο Μπεζιέ και σε αυτό πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων οι εγκαταστάσεις λειτουργούν ικανοποιητικά. Ευχαριστώ. Κάποιος κανείς θέλει να πάρει το λόγο. Ο συνάδελφος. Ευχαριστώ. Δεν ξεκίνησα από την αρχή την παρακολούθηση, αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα της Κομισιόν είναι λίγο βεβαιασμένο. Λέει ότι το δικαίωμα, το δικαίωμα θα πρέπει να ισχύσει και η η γαλλική νομοθεσία είναι αυστηρή ούτως ή άλλως αυτό το θέμα. Αλλά εγώ ρωτάω, δόθηκε η σε αυτο το θεμα αλλα εγω ρωταω δοθηκε Η μελέτη επιπτώσεων δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία ζημία, καμία βλάβη. Ε, ποιο είναι το αποτέλεσμα της μελέτης επιπτώσεων. Με ποιο τρόπο ε, εξαφανίζονται τα απόβλητα αφού συλλεγούν τα λύματα. Ε, μιλάμε τώρα για διάφορε λεπτομέρειε οι οποίες δεν μα έχουν δοθεί. δεν είχα αρκετό χρόνο να τα, κοιτάξω, να τα κοιτάξω αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα εστιάζουν στη γαλλική νομοθεσία. Δεν δίνουν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα. Ούτως ώστε να διαμορφώσουμε κι εμείς γνώμη. Ε, Συμφωνώ με αυτή την παρατήρηση η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ικανοποιητική. Συνδυάζει, την, μάλλον συνδέει και εξαρτάται την απάντησή της από την απάντηση των γαλλικών αρχών. Οι οποίες αρχές είπαν ότι θα αλλάξουν το σύστημα συλλογής λιμάτων. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί και ότι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή λοιπόν. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να πιέσουμε τις τοπικές αρχές για να ανταποκριθούν πάρα αυτά ε, στα αιτήματα των πολιτών και στα, στις ανησυχίες, και να απαντήσουν στις ανησυχίες των πολιτών. Θα στείλουμε ένα επίσημο, μια, μια επίσημη επιστολή στις τοπικές αρχές για να τους ζητήσουμε να παρέμβουν και να μας πούν μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα σκοπεύουν να παρέμβουν όπως έχουν ανακοινώσει. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουν οι συνάδελφοι να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ε, το ζήτημα με βάση τις αρμοδιότητές της. Πιστεύω ότι δεν υπήρξε αυτήν την περίπτωση πραγματικός έλεγχος. Απλώς σημειώνει την κατάσταση όπως έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν νομίζω ότι είναι καλύτερη συμπεριφορά αυτή. Επομένως παραμένει ανοιχτή η αναφορά και Τώρα περνάω στο σημείο 18. Θα δώσω το λόγο στον αναφέροντα, τον κύριο Χάκανσον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου ζητήσατε να... που μου επιτρέψατε μάλλον να παρουσιάσω αυτή την αναφορά. Είμαστε μια οργάνωση 100% ε, ιδιωτική, 135.000 μέλη. Ε, μιλώ εξ ονόματος του Διευθυντή σήμερα. Εγώ ασχολούμαι ε, με θέματα ε, υδάτινης πολιτικής. Μιλάμε για την ε, βυθοκόρηση με σκοπό τη συγκομιδή μυδιών σε περιοχέ του δικτύου Natura 2000. Αυτό επηρεάζει τη θαλάσσια ζωή ε, μια περιοχή η οποία πρέπει να προστατευτεί. Νομίζω ότι παραβιάζουμε τα άρθρα 6.2 και 6.3 της ε, οδηγίας για τους οικότοπους. Γι' αυτό εμείς λοιπόν ε, μέσα στην αδυναμία μας στραφήκαμε προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταπολεμηθούν οι άδειε ε, που δόθηκαν Εμεί δεν είμαστε κατά τη μυδοκαλλιέργεια σε καμία περίπτωση, αν αυτή γίνεται με βιώσιμο τρόπο. Η χθιοκαλλιέργεια είναι μια βιώσιμη δραστηριότητα στην βυθοκόρηση ε, και τη συγκομιδή μυδιών μέσω βυθοκόρηση, που αντίθετα αυτή είναι μια καταστροφική δραστηριότητα. Το 2008 ε, αρχίσαν να γεννιόνται αμφιβολίε, γι' αυτό στραφήκαμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν ξέρουμε αν γίνεται σωστή παρακολούθηση Υπάρχει μια απόφαση του ΔΕΚ, το οποίο έλεγε ότι θα πρέπει να αποδειχθεί με τρόπο αναμφίβολο ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα, οικονομική δραστηριότητα, δεν επηρεάζει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Δεν, ξέρω αν ε, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη από τους υπευθύνους. Και εγώ πιστεύω ότι στην πραγματικότητα καταστρέφουμε αυτά τα, αυτούς τους χώρους που υποτίθεται ότι προστατεύουμε μέσω την, α, της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε επιστημονικά στοιχεία τα οποία πρέπει να μας δοθούν καταρχάς και μετά θα πρέπει να τα σεβαστούν οι αρμόδιες αρχές. Δεν νομίζω ότι αυτό γίνεται στη Δανία. Αντίθετα, λαμβάνονται λανθασμένες αποφάσεις, ε, έχουμε ανελειπή ε, επιστημονικά στοιχεία, δεν κάνουμε αυτά που μας ε, επιτρέπουν οι περιβαλλοντικές οδηγίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε απευθυνθεί στις τοπικές αρχές, έχουμε ένα συνεχή διάλογο με το Υπουργείο, αλλά δεν έχουμε πετύχει αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ήρθαμε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό στείλαμε ένα φορά στην Επιτροπή σας. Οι αναφέροντες πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη διαχείριση των δικτύων της Natura 2000 στη Δανία, συμμορφώνονται με την οδηγία για τους οικότοπους, την οδηγία Habitat, ειδικά σε ό,τι αφορά την βυθοκόρηση με σκοπό τη συγκομιδή ιδιών. Ε, χαίρομαι που η Κομισιόν παίρνει το παράπονό μας και το πρόβλημά μας πολύ θα σοβαρά και έχει στείλει τον Οκτώβριο του 2010 επίσημη επιστολή στην Δανία. Επίσης χαίρομαι που η Επιτροπή σας έχει βάλει το θέμα αυτό στη σημερινή μερίσια διάταξη. Το γεγονός και μόνο ότι τέθηκε αυτό το θέμα ε, είναι θετικό. Το 2008 ελέγχθη ότι οι άδειε αυτές, αν εκδοθούν, θα έχουν ε, επιζήμες επιπτώσεις. Ε, το 2009 και 2010 ε, βελτιώθηκε η κατάσταση. Οι νέες, ε, τα νέα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι η διθοκόρηση είναι πάρα πολύ προβληματική διαδικασία και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παρά τις μελέτες όμως επιπτώσεων που, είναι, που δείχνουν ότι είναι προβληματική αυτή η δραστηριότητα. Ε, η βυθοκόρηση συνεχίστηκε και το 2009 και 2010. Και τώρα οι περιοχές αυτές ε, πλήττονται περιβαλλοντικά και η Δανία δεν σέβεται τις υποχρεώσεις της. Η Δανέζικη κυβέρνηση λοιπόν λέει τώρα ότι δεν υπάρχουν τελικοί δεν υπάρχουν στόχοι, ας πούμε, τελικοί για τους χώρους του δικτύου Natura 2000. Αυτό όμως είναι σε αντίθεση με το άρθρο 6 της ε, σχετικής οδηγίας. Η κυβέρνηση λέει επίσης ότι η βυθοκόρηση για τη συγκομιδή ημιδιών ε, χρειάζεται και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη βυθοκόρηση. Αλλά αυτά δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα όταν μιλάμε για την, προστα... περιβαλλοντική προστασία αυτών των περιοχών. Οι Δανέζικες αρχές επίσης προσπαθεί να πει ότι Υπάρχουν ενδυνάμει απειλέ στου χώρου ε, του Natura 2000. Η πρώτο διακόπτει τον ομιλητή λέγοντα ότι τελείωσε ο χρόνο του. Από πλευρά τη Επιτροπή. Σουζάν Βέγκερφελντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε όπως σας είπα ξεκίνησε η περίπτωση αυτή το 2008 με ε, την ε, αναφορά της ε, Δανικής οργάνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και οι αρχές του, της Δανίας ε, συνέχισαν να επιτρέπουν την βυθοκόρηση αυτή για την ε, συγκομιδή μηδιών το 2009 και 2010. Ε, βέβαια, η, ε, ε, η μελέτη δεν συνείδε με τις ε, οι υποχρεώσεις που καθορίζει η σχετική νομοθεσία και υπήρχαν κενά. Από ό,τι ε, ενημερωθήκαμε και σε άλλες περιπτώσεις σήμερα η διάταξη 6 για τα οικοσυστήματα προβλέπει ε, να υπάρχει μία μελέτη σκοπιμότητος για την επιρροή σε χώρους που διέπονται από το πρόγραμμα Natura 2000 και αυτό έχει σχέση με την χωρίζηση ή όχι της αδείας υλοποιήσεως του προγράμματος. Τα επιχειρήματα αυτά απευθύνθηκαν στην Δανία, στις δανεικές αρχές ε, και ζητήσαμε πληροφορίες όπως είπαμε ε, ή στην Επιτροπή ήδη το 2009. Το 2010 η Επιτροπή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η αδειοδότηση ε, αφήνει ερωτηματικά διότι φαίνεται ότι η αξιολόγηση ε, των επιπτώσεων επί της αλληλείας, επί των συσσωρευτικών επιπτώσεων με ε, την ε, διατήρηση των τόπων και την συνεκτίμηση της καλύτερης διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αξιολογήσεις αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 και δεν έπρεπε να έχει εγκριθεί η βυθοκόρηση για την ε, συγκομιδή ε, μηδιών στην, ε, στις 28 Οκτωβρίου πέρυσι η Επιτροπή ε, απεφάσισε να αποστείλει ε, η προειδοποιητική επιστολή στη Δανία σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης της, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η Δανία απάντησε και αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την απάντηση. Ευχαριστώ λέει η κυρία Όκεν. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το γεγονός ότι έφτασε η υπόθεση αυτή στην Επιτροπή μας, γιατί εμείς έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Το ανοιχτό πνεύμα είναι προϋπόθεση. Είναι προϋπόθεση για να συμμετάσχουν οι πολίτες στις διαδικασίες. Και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος χρειάζεται την εμπλοκή των πολιτών. Πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες για τα διαμοιβόμενα και διακυβευόμενα. Στη Δανία έχουμε το εξή πρόβλημα. Η δανέζικη κυβέρνηση πιστεύει ότι είναι καλύτερη από οποιονδήποτε άλλο. Έχουμε την αίσθηση ότι προστατεύουμε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο το περιβάλλον και ότι στην υπέροχη Δανία τίποτα δεν πάει στραβά. Τίποτα δεν πάει στραβά στο βασίλειο τη Δανία. Αλλά κάτι δεν πάει καλά με αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ρωτήσουμε την Κομισιόν. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να, έχουμε, να λάβουμε πλήρη γνώση της επιστολής που στείλατε και της απάντησης της κυβέρνησης. Έχω την αίσθηση ότι όλα τα προβλήματα από αυτό απορρέουν. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η φύση της δανέζικης κυβέρνησης και νομίζω ότι η δανέζικη κυβέρνηση απλώς επιτρέπει να συμβούν αυτά που καταλογίζουμε εδώ αν σεβόμασταν την ε, διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σύμβαση Όρχους, όλες αυτές τις συμβάσεις και αρχές και, και κείμενα που έχουμε, ε, τότε γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε γνώση και για τα έγγραφα τα οποία ανταλλάξετε μεταξύ σας. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτές τις διαδικασίες και κλεισμένων των θυρών. Εγώ έχω συνεργαστεί με τέτοιες οργανώσεις πολύ συχνά. Το πρόβλημα είναι ότι ε, σπάμε τα μούτρα μας πάνω στις κλειστές πόρτες. Ε, υπάρχουν και άλλα δίκτυα του Natura 2000 όπου γίνεται διθοκόρηση για τη συγκομιδή ιδιών και όλες αυτές οι περιοχές καλύπτονται από αυτή την αίτηση. Ο κ. Μποστινάρου. Πρώτο, πρώτο. Αυτή τη φορά με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενήργησε ορθά και πέρασε το μήνυμα στην κυβέρνηση της Δανίας. Επομένως, νομίζω ότι η αναφορά θα πρέπει να μείνει ανοιχτή έως ότου επιληθεί το πρόβλημα. Όμως, όμως, εν κατακλείδη να σας πω ως ακροτρέφτε παρατηρήσει ότι έχουμε εδώ πέρα έλλειψη διαφάνειας γιατί δεν μιλούμε για πνευματική ιδιοκτησία εν προκειμένου ούτε για σχεδιασμό όπλων υψηλής τεχνολογίας. Απλώς εδώ πρόκειται για κάτι που είναι φυσιολογικό το οποίο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους. Και γι' αυτό σας λέω, δεν καταλαβαίνω την κυβέρνηση της Δανίας η οποία ακολουθεί την οδό της μυστικότητας που είναι τόσο καταστροφικό για το κύρος της. Έχω δύο σύντομες ε, παρατηρήσεις. Καταρχήν ε, θα πρέπει το θέμα να παραμείνει ανοιχτό που να υπάρξει τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεύτερον, μία έλλειψη διαφάνειας δημιουργεί και δυσπιστία και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρχει διότι ε, πρέπει να κοιτάξουμε να μειώσουμε τη δυσπιστία ε, διότι ε, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε στο τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία φαίνεται να έχει λάβει τα ενδεικνυόμενα μέσα για να δούμε πώς θα ε, γνωρίζουμε καλύτερα το τι συμβαίνει όσον αφορά τα στοιχεία ε, ξέρω ότι στην σοσιαλιστική εποχή αποκρύπτονται τέτοια στοιχεία αλλά τώρα αντιλαμβάνουμε ότι είναι ανοιχτά και προσβάσιμα. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απαντήσει και θα του δώσω το λόγο. Τον παρακαλώ να απαντήσει στα ερωτήματα των συναδέλφων και να μας δώσει πρόσβαση στα κείμενα που ζητάμε, σε επιστολές εν προκειμένου, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε γνώση. Έχετε το λόγο. Λέγομαι Λίν Κάσμιν. Δουλεύω στην νομική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το χειρισμό των υποθέσεων παράβασης που ανέφερε στην αδελφό μου. Σε ό,τι αφορά την ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας ε, στις ανταλλαγές επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Δανίας. Η Κομισιόν ε, είναι δεσμευμένη από τους όρους του καονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2001 είναι ο κανονισμός 1049 ε, του 2001. Και με βάση τους όρους αυτού του κανονισμού η Κομισιόν καταρχήν δίνει άξις, ε, πρόσβαση στα έγγραφα κατόπιν αιτήματος. Αλλά αυτή η γενική, ε, αυτή η γενική διάταξη έχει διάφορες εξαιρέσεις. Μία από αυτές αφορά την περίπτωση όπου η Κομισιόν εμπλέκεται σε μια διαδικασία παράβασης ή έρευνας με ένα κράτος μέλος. Το δικαστήριο, το ΒΕΚ, αποφάσισε ότι η Κομισιόν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να λάβει υπόψη τη δυνατότητα επίλυσης με φιλικό τρόπο ε, του θέματος αυτού, α, εφόσον το θέλει το κράτος μέλος. Επομένως, η Κομισιόν σε αυτή την περίπτωση δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει έγγραφα τα οποία συνδέονται με μια συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κράτους μέλους. Ε, δεσμευόμαστε από τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό που μπορώ να πω είναι, αυτή τη στιγμή η διαφορά ολοκληρωθεί, τότε η Κομισιόν θα δώσει στο κοινό, σε εσά εμπροκειμένου, όλα τα έγγραφα ε, τα σχετικά με την ε, Δανία. Πρέπει όμως να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για τη διαφορά Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δανίας. Κυρία Όκεν, δεν θέλω να ανοίξετε αυτή τη συζήτηση. Μία σύντομη απάντηση, μια διευκρίνηση, σας παρακαλώ. Η απάντηση της κυρίας Όκεν χωρίς μικρόφωνο. Απλά κάτι να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει κυρία Όκεν. Εάν αποδεχθεί η κυβέρνηση της Δανίας το να υπάρχει πρόσβαση και αν θεωρηθεί ότι όλα καλά και εσείς συμφωνείτε ότι όλα καλά, το λέω γιατί τα επιχειρήματα τα οποία προτάξατε ήταν αυτό, ότι εάν αυτοί δεχθούν, νο, έχουμε ανοιχτή κοινωνία, έχουμε τέτοιου είδους παράδοση, κουλτούρα, διαφάνειας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας και το, το όρχος στο οποίο βγήκε η σύμβαση είναι η πόλη μας είμαστε περήφανοι γι' αυτό επομένως τι λέτε Una risposta. Ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ανοιχτή πρόσβαση σήμερα και αυτό είναι και το πρόβλημα. Εάν τώρα η δανεική κυβέρνηση ισχυριστεί ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται να είναι πρόσβαση, τα έγγραφα, τότε εμεί θα το, το κοιτάξουμε, θα το μελετήσουμε και θα σα πούμε. Πολύ ωραία, συγκεκριμένη απάντηση. Ένα λεπτό για την απάντηση που θα δώσουν οι αναφέροντε τώρα. Κοιτάξτε. Θα πρέπει να δούμε πώς είπε η κυρία Άουγεν. Να δούμε κατά πόσο αυτό γίνεται και αλλού στη χώρα. Έχουμε και άλλες περιοχές του Natura 2000 όπου συντρέχει η ίδια κατάσταση και να δούμε κατά πόσο εκεί πέρα θα υπάρξουν και στο μέλλον άλλες αδειοδοτήσεις. Μας τα είπε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει τελικά πολιτική βούληση, βούληση ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον. Και έτσι να ισχύσει η, η εθνική νομοθεσία παντού Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την εξέλιξη υπόθεσης, να υπάρξει διαφάνεια, να ληφθεί η σωστή απόφαση. Και αυτό ενδεχομένως συνδεστεί και με απόφαση του Ευρωπαϊκού Επιδεστηρίου το οποίο θα υποχρεώσει την, Ευρωπαϊκή την Δανέζικη κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της αναφοράς. Η αναφορά παραμένει ανοιχτή, όπως ζήτησαν και οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο. Ούτως ή άλλως περιμένουμε απαντήσεις. Και θα διαβάσουμε κάπου αν, για τη στάση της δανέζικης κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ όλους. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 19, για μια αποστολή που έγινε στην Αυστρία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίλαντ για να μας παρουσιάσει συνοπτικά το θέμα αυτό. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να υποφεληθώ από την επανεξέταση του θέματος στο να τονίσουμε ότι δεν θα έπρεπε να συμμετέχουμε σε τέτοιες καταστάσεις διότι εδώ μιλάμε για μία αναφορά του 2007 που ξεκίνησε του 2007 και χρειάστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2008 για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία επεξεργαστήκαμε πλέον το φινόπορο οπότε από πλευράς

Ε, από πλευράς αξιολογήσεως δεν μπορέσαμε να, το, την, ε, ε, να την κάνουμε πριν από το καλοκαίρι του επομένου έτους και βλέπουμε ότι αυτή η καθυστέρηση δεν λήφθηκε υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, όταν για την συγκέντρωση στοιχείων δεν μπορούμε παρά να πάμε καλοκαίρι θα έπρεπε η διερευνητική ε, επίσης και οι της να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ο ανώτατος δικαστής για εθνικές υποθέσεις ε, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι οριακές τιμές και η αξιολόγησή τους. Δηλαδή, από ποιο σημείο και πέρα χρειάζεται υποχρεωτικά μία μελέτη αξιολογήσεως των επιπτώσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είπε ότι αυτές οι οριακές τιμές θα πρέπει να εξεταστούν ε, περιοριστικά. Συνήθως λέγεται ότι εάν πρόκειται για ένα λεπτό θέμα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μελέτη των επιπτώσεων αλλά εάν το πρόγραμμα έχει μία συγκεκριμένη μεγάλη έκταση τότε πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ένα τέτοιο επίπεδο. Τότε ε, σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο η έκταση της περιοχής ήταν 20 εκτάρια έκτοτε μειώθηκε στα 10 εκτάρια. Τώρα όμως έχουμε υπερβεί τα 10 εκτάρια και τότε οι αρχές και οι εργολήπτες πίστευαν ότι δεν είχαν υπερβεί το κατώτατο όριο εφόσον πρόκειται περίπου για 18 εκτάρια. Πήγαμε λοιπόν και επισκεφθήκαμε την περιοχή για να αξιολογήσουμε την κατάσταση και συγχρόνως να μπορέσουμε να έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερομένους για να δούμε αν ήταν ένα θέμα το οποίο είχε σε σχέση με την έκταση ή όχι γιατί ε, πιστεύω ότι σε αυτό βοήθησε η οχι γιατι πιστευω οτι σε αυτο βοηθησε η επίσκεψη καθότι εγώ πριν την επίσκεψη δεν ήμουνα σε θέση να σκεφτώ ότι έπρεπε κανείς να λάβει υπόψη και τα πάρκινγκ ε, και ουσιαστικά φαίνεται ότι εις ε, το χαμηλότερο επίπεδο ε, του σκι στο Μελάου ε, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων μειώθηκε δηλαδή οι διαστάσεις των δυνατοτήτων παρκαρίσματος ε, δεν χρησιμοποιόντουσαν πλέον ε, και είχαν ενσωματωθεί οι δυνατότητες σταθμεύσεως και συμπεριληφθεί για τους επισκέπτες που θα προστίθεντα και ε, υπάρχει μια μεγάλη ε, έκταση όσον αφορά ε, το χώρο σταθμεύσεως που δεν είχε αρχικά περιληφθεί εις τους υπολογισμούς. Τώρα, το εάν είναι ευαίσθητο το, ευαίσθητος ο χώρος ώστε να χρειαστεί μία μελέτη Τη της σκοπιμότητος της περιοχής είναι κάτι που είναι ακόμη αμφιλεγόμενο διότι εμείς βασιστήκαμε στις αξιολογήσεις των αρχών μπορεί να έχει κανείς ε, μία πιο θετική αξιολόγηση ή μία πιο αρνητική και πιστεύω ότι γενικά τα κράτη-μέρη πρέπει να εξαντλήσουν τις δυνατότητες όστε ώστε να παρουσιάζουν αποτελέσματα τα οποία μπορούν να ε, ε, τύχουν μίας δικαστικής αξιολογήσεως. Στο σημείο όμως αυτό βρισκόμαστε σε ε, οριακό σημείο όσον αφορά τις αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Εμείς δεν είμαστε ανώτατο δικαστήριο και στο οικοδομικό δίκαιο υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι συνυπολογίζονται και ε, είναι δύσκολο να προβούμε οι συμπεράσματα. Ε, είναι όμως ε, σε ένα τομέα όπου πρέπει να κοιτάξουμε και στις οικονομικές πτυχές και τις δυνατότητες εκμεταλλεύσεως για τον εντόπιο πληθυσμό. Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα στο τομέα αυτό διότι εκεί ε, σε αυτή την περιοχή υπάρχουν διάφορα κίνητρα δηλαδή στο Μέλαου μειώθηκαν οι διανυκτερεύσεις ε, και ε, στο Ντάμιλς αυξήθηκαν και άρα το Μέλαου ήθελε να συμπεριληφθεί στην περιοχή γι' αυτό και ήταν πιο συγκρατημένοι οι κάτοικοι παρόλο που δεν ήταν ενθουσιασμένοι με τις εξελίξεις. Άπαξ όμως και ε, ε, ε, ασχολεί, συμπεριελήφθη στην αξιολόγηση και ο χώρος ξενοδοχείων τότε θεωρήθηκε ότι άπαξ και θα υπήρχαν δυνατότητες περισσότερων διανυκτερεύσεων και περισσότερων ενδιαφερομένων τότε είπαν ότι έπρεπε να διευρυνθεί και ο σκόρος σκι και ο η χιονοδρομική ζώνη και θα έπρεπε ε, να δούμε ε, αν ε, προσετέθησαν χώροι 1,5 εκταρίου ώστε όντως να υπερβούμε το κατώτατο όριο του αυστριακού δικαίου των 20 εκταρίων. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, αντικρώμενες σε αυτό και πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε μία χώρα όπου καλό θα ήταν να δούμε πώς ε, θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν δύο νευραλγικά σημεία ε, που πρέπει να αξιολογήσουμε. Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποφασίσουμε τελεσίδικα δύο, όπως είπα, ουσιαστικά θέματα. Καταρχήν πρέπει να δούμε ε, στην περίπτωση του Ντάμιλς αν ε, σύμφωνα με την εθνική ε, νομοθεσία υπάρχει μία υπέρβαση του ισχύοντος κατώτατου ορίου δηλαδή αν η ευρωπαϊκή αξιολόγηση είναι σωστή διότι μπορούμε να δούμε αν υπάρχει μία ενεργειακή εγκατάσταση όπου παράγεται αέριο και θέρμανση και τα δύο επίπεδα χωριστά είναι κάτω από το κατώτατο όριο τότε μπορεί κανείς ε, να είναι επινοητικός και ακόμη και σε αυτές τις χιονοδρομικές περιοχές μπορεί κανείς ε, να διαχωρίσει τα διάφορα ε, επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνυπολογιστεί. Αλλά η δυνατότητα διαχωρισμού των προγραμμάτων γνωρίζουμε ακριβώς ε, ποιες είναι οι ευρωπαϊκές επιταγές για το 2011 και πρέπει να δούμε εάν η αυστριακή πλευρά έχει συμμορφωθεί με αυτές τις επιταγές και δεύτερον πρέπει να δούμε εάν οι χιονοδρομικές πίστες, η συνολική επιφάνεια μιας χιονοδρομικής πίστας μπορεί να αποκλειστεί από, την, από το πρόγραμμα και τον συνυπολογισμό διότι οι αυστριακές αρχές είπαν ότι όπου δεν υπάρχουν αραγές στην τοπογραφία τότε ε, εξαιρεί περιοχές αυτές. Ε, υπάρχει λοιπόν παρεμφερές ε, περιστατικό και σε άλλες χώρες και καλό θα ήταν να γίνει μία προφορική επερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα η κυρία Μάριαν Μίλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Έκανε από το 2007 αυτή αναφορά και για να μπορέσουμε να καταλούμε καλύτερα πώς έχει η κατάσταση θα πρέπει να δούμε λίγο την ε, προϊστορία, το ιστορικό πλαίσιο αυτού του θέματος. Όντως έχουμε εδώ πέρα ε, την οδηγία της ε, Μέλης επιπτώσεων που και ορίζει ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη διακρατική ευχαίρεια για τα έργα του δευτέρου παραδείγματος όπως το συγκεκριμένο έργο, πρόγραμμα και επομένως διακριτήριος ευχαίρεια των κατομελών είναι είτε περιτοσιολογικά να εξετάζουν κάθε έργο το οποίο εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση και έτσι να υπάρχει κάποια προκαταρκτική αξιολόγηση του αν υπάρχουν επιπτώσεις του περιβάλλον ή επίσης μπορεί, είναι δυνατόν έτσι να έχουμε κάποια κριτήρια, ε, κάποια κατόφλια σε σχέση με το να κριθεί ποια προγράμματα πρέπει να περάσουν από μελέτη αξιολόγηση. Μπορούν το πάντως να συνδυάσουν την πρώτη και δεύτερη εκδοχή. Το 2007 η αστρική νομοθεσία είχε τα 20 εκτάρια ως κατόφλια και ανεφέρετο ότι μόνο σε περίπτωση που έχουμε επιφάνεια 20 εκατομμύρια και άνω. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επομένως, οτιδήποτε κάτω από αυτό το εμβαδόν του κατοφλίου απαλλάσσεται τις υποχρεώσεις και έτσι είχε η κατάσταση. Κάτω των χρόνων αφήξεως τέλο πάντων υποβολή τη αναφοράς και υπ' αυτού του όρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τις ε, επαφέ με τις αυστριακέ αρχές. Εξήγησε δε ότι η νομοθεσία αυτή δεν συμβαδίζει με την κείμενη νομοθεσία αλλά και με τις αποφάσεις και την ομολογία του ΔΕΚ. Αυτό έγινε αποδεκτό ως επιχείρημα από την Αυστρία, η οποία τροποποίησε την εφαρμοστική της νομοθεσία και διάλεξε την συνδυασμένη προσέγγιση σε σχέση με το κατόφλι, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υποχρέωσε το να ελέγχεται το αν συντρέχει περίπτωση κατοφλίου εκ των προτέρων. Βέβαια, το τωρινό κατόφλι είναι διαφορετικό από το κατόφλι που είχε το 2007. Είχαμε τα 20 εκτάρια τώρα, όμως ο κανόνας στην νομοθεσία, ο κανόνας δεν είναι ότι μόνο ότι είναι πιο μεγάλο από μια τέτοια επιφάνεια που να περάσει από μελέτη επιπτώσεων. Και άρα ότι όλα κάτω από 20 εκτάρια απαράσσονται τις υποχρεώσεις. Αυτό που ισχύει σημαίνει ότι οποιοδήποτε έργο που καλύπτει φάνη πάνω από 20 εκτάρια θα πρέπει να περάσει από μελέτη επιπτώσεων. Την άλλη μεριά, τα έργα τα οποία δεν φτάνουν σε επιφάνεια μέχρι αυτό το κατόφλι θα πρέπει να υποστούν μια εξέταση του, του τι ισχύει όσον αφορά τη μελέτη των επιπτώσεων και άρα δεν απαλλάσσονται αυτοδικαίως. Να, ποια ήταν η αλλαγή που έγινε στην Αυστριακή νομοθεσία το 2009. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σύμφωνο με την οδηγία για τη μελέτη των επιπτώσεων. Επομένως, θεωρήθηκε ότι το εν λόγω έργο Καλή επιφάνεια κάτω από 20 εκτάρια και επομένως γι' αυτό και έγινε αυτό ο έλεγχο του, του screening. Οπότε και οι κατέληξαν στο ότι το έργο δεν θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. επομένω και από διαδικαστική και οικονομικής πλευρά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ στηρίξει περίπτωση παραβίασης της οδηγίας για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενημερωθήκαμε από την Αυστρία για την εξέλιξη της διαδικασίας και εμείς ενημερώσαμε Έχουμε τώρα κάποιους ε, επίσης ανεξάρτητους εμπειρογνώμους οι οποίοι έχουν εμπλακεί στη δουλειά. Το δε τελικό αποτέλεσμα επίσης έγινε αποδεκτό από τον από κάποιον τέλος πάντων ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο για τα θέματα περιβάλλοντος. Τώρα, αυτό το οποίο προκύπτει από αυτή την προβληματική είναι βέβαια ότι κομβική σημασία έχει εδώ πέρα το κατόφλι το οποίο έχει οριστεί από την Αυστριακή νομοθεσία γιατί αυτό είναι ένα εύκολο, εφαρμόσιμο, αντικειμενικό κριτήριο. Εάν πληρούνται οι όροι του κατοφλίου, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το αν πρέπει ή όχι να γίνει μελέτη επιπτώσεων. Όμως, οδηγία δεν ορίζει με λεπτομέρειες για το πώς τα κράτη-μέλη ορίζουν το κατόφλι. και το κατόφλι το οποίο αφορά την ε, επιφάνεια του εδάφους επί της οποίας εκτελείται το έργο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι, είναι, ότι αυτό ταυτίζεται και με την επιφάνεια, με το εμβαδόν, με, με, με το χώρο όπου υπάρχουν επισημαίνουν οι επιπτώσεις οι περιβαλλοντικές και επομένως πρέπει να εξεταστεί αυτό και όπως θα πρέπει να εξεταστεί και με το screening το τι είδους περιβαλλοντικές συνέπειες έχουμε εκεί που γίνεται το έργο, σε εκείνη την περιοχή. Έχουμε κάποιες αναθεντήριες γραμμές για το πώς γίνεται αυτό το screening. Αυτές ε, το 2001 και έχουμε τώρα και κάποιες άλλες συνέπειες που συντρέχουν σωρευτικά. Ας πούμε για την κίνηση, την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και άλλα φαινόμενα που είναι εκτός του κυρίως χώρου εκτέλεσης του έργου, οπότε δεν είναι δυνατόν θέλουμε να πούμε ότι το screening και αυτός ο έλεγχος θα περιορίζεται μόνο στην περιοχή επιφάνεια εκτέλεσης του έργου. Ευχαριστούμε κύριε Λότερ Πέτερ. Πρώτα απ' όλους ο αναφέρον. Άλλος είναι. Έτσι δεν είναι. Σε ότιμες κυρίες και κύριοι της Επιτροπής Αναφορών ορισμένες ανέπαφες ε, περιοχές φυσικού κάλους ε, αποτελούν εξαίρεση στην Ευρώπη και ο χειμερινός τουρισμός επεκτείνεται όλο και περισσότερο και ιδίως στο Φοράντελμπερκ στην ε, Αυστρία που έχει την μεγαλύτερη πυκνότητα χιονοδρομικών σταθμών και με το συνδυασμό του Ντάμιλς και του Μέλαου ε, υπήρξε μία επέκταση της χιονοδρομικής ζώνης η οποία προκάλεσε μεγάλες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια ε, υπήρξαν ε, συνεχείς επικεφαλίδες στον τύπο σχετικά με το θέμα αυτό και η Επιτροπή Δράσεως δεν γνωρίζει καμία άλλη χιονοδρομική περιοχή που να έχει καταστραφεί ε, τόσο ποσοστό της ε, φυσικής περιοχής ε, όσο στην περιοχή Ντάμιλ Σμέλαου και πουθενά αλλού δεν έχουν υπάρξει αυτά τα αποτελέσματα για να μπορέσουν να συνδυαστούν τα χιονοδρομικά κέντρα Ντάμιλς Ντάμιλς-Μέλαου χρειάστηκαν αυτές οι επιπτώσεις ε, υπήρξαν σημαντικές επεμβάσεις και στους βιοτόπους και ε, τελικώς όλα αυτά ε, ε, παραπέμφθηκαν ή στις αρμόδιες αρχές η οποία θεώρησε ότι δεν χρειάζεται μία περιβαλλοντολογική μελέτη. Γι' αυτό και το 2007 υποβάλαμε την αναφορά στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας ε, ε, ε, διαδικασίες αδειοδοτήσεως να εξεταστούν διότι υπήρχαν κραυγαλές παραβιάσεις των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της σχετικής οδηγίας. Υπήρχαν λοιπόν πολλές περιβαλλοντολογικές οργανώσεις στην Αυστρία, η Ένωση στη Βιέννη και η Ένωση της Προστατεύσεως των η ε, Ένωση ε, για τη φύση του Φοράντελμπεργκ ε, όλοι συσπυρώθηκαν αλλά παρόλη την αναφορά δεν έγινε μία περιβαλλοντολογική μελέτη παρόλο που είχαν υπερβεί οι εγκαταστάσεις στο κατώτατο όριο των 20 εκταρίων διότι βλέπουμε ότι ήδη η ελάχιστη περιοχή ήταν 18,5 εκτάρια ε, και χρειάζεται επιπλέον ε, ένας, ε, μία λίμνη για την παραγωγή τεχνητού χιονιού. Άρα υπήρχε ε, μια υπέρβαση του κατωτάτου ορίου και θα έπρεπε σύμφωνα με την νέα οδηγία ε, να ε, θεωρήσει κανείς ότι τα κατώτερα όρια σαφώς έχουν υπερβεί. Με, τις, με τον νέο χιονοδρομικό αναβατήρα μάλιστα χρειαζόταν να γίνει οπωσδήποτε μια νέα μελέτη διότι διορθώθηκε και το συνολικό περιβάλλον, δηλαδή για να υπάρχει περισσότερος χώρος ε, για τον αναβατήρα αυτό ε, επενέβησαν εις ε, το, εις έδαφος και θα χρειαστούν και στο μέλλον διορθωτικές κινήσεις. Αυτά τα στοιχεία έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Αναφορών και έκτοτε έχουμε και μία τοποθέτηση ενός καθηγητού πανεπιστημίου επί του θέματος διότι πρόκειται για έναν ε, διεθνώς γνωστό εμπειρογνώμονα ο οποίος διαβλέπει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις από ό,τι διαπίστωσε η ε, επίσκεψη της ε, αντιπροσωπείας της αρχές του Σεπτεμβρίου το 2010. Από βιολογικής πλευράς υπήρξε μια σημαντική επιδίνωση και σε μια περιοχή ε, είδαμε ότι κατεστράφει ε, ένας μεγάλος χώρος ε, για να μπορέσουν να συνδυαστούν οι χιονοδρομικές περιοχές. Πρέπει να υπάρξει ε, μία αντικειμενική αξιολόγηση και ελπίζουμε ότι η απόφασή σας για το Φοράντελμπεργκ θα μπορέσει να επηρεάσει ε, και την νομιμότητα των επομένων εγχειρημάτων ε, και ε, σας έχουμε επισυνάψει και διάφορες φωτογραφίες τις οποίες μπορείτε να αξιολογήσετε. Ευχαριστώ κύριος Λίχτεμπεργκ. Ευχαριστώ. Όντω είχα συμμετάσχει σε αυτήν ε, την ε, μικρή αντιπροσωπεία η οποία μετέβη στην Αυστρία για να εξετάσει επιτόπου την ε, κατάσταση. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ήταν και εδώ δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες που ανέφερε ο συνάδελφος αλλά γενικώ αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ήταν ότι αυτό που θεωρούσαμε σαν οδηγία ε, ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δηλαδή, εξηγώ, υπάρχει μία χιονοδρομική ζώνη χωρίς να περιλαμβάνουμε τις πίστες. Δηλαδή, δεν ξεκινάμε από τα τρία τετραγωνικά που χρειάζεται να εδράσει το, ο αναβατήρας ή όπου χρειάζεται να εδράσουν ε, οι φωτισμοί, αλλά ξεκινάμε μόνο από την πίστα που θα πρέπει να χιονιστεί. Και υπάρχουν ε, παρελκόμενες επιπτώσεις διότι το σήμερα χρησιμοποιεί κανείς και το ε, χιονοδρομικό χώρο εκτός πίστας. Οπότε, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά το screening έπρεπε να μην έχει κανείς περιοριστεί εις τον έλεγχο των περιοχών που τροποποιήθηκαν όσον αφορά το βασικό έδαφος αλλά πολύ πιο ευρέως έπρεπε να έχουμε βασίσει την μελέτη αξιολογήσεως. Αυτό θα ήταν η σωστή ερμηνεία και η ερμηνεία η οποία έγινε όπως ελέγχθηκε προηγουμένως αναφερόταν μόνο στην επαλήθευση του κατωτέρου τα του ορίου, αν είμαστε πάνω ή κάτω από τα 20 εκτάρια. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι θέμα γενικής αξιολόγησης και έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Το 2003 υπήρξε μία μελέτη από την εταιρεία κατασκευή των αναβατήρων που παρουσίασε το ολικό εγχείρημα το οποίο ε, θα περιλαμβανόταν. Αλλά αυτό το οποίο μας έδωσαν δεν ήταν το ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο βαθμιαία επεκτείνεται και ξεπερνά πλήρως ε, το ε, ε, την οδηγία ΕΠΕ. Δηλαδή χρειάζεται να υπάρξει μία συνολική αξιολόγηση η οποία δεν έχει γίνει και αυτό για μας είναι ένα πολύ βασικό σημείο διότι διαφορετικά με αυτή την ε, στρατηγική σαλαμοποίησεως δηλαδή την κατάτμιση των προγραμμάτων σε μικρότερες περιοχές ε, θα επιτρέψει στα κράτη να παρακάμψουν την οδηγία αυτή. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να θίξουμε εδώ διότι δεν ερμηνεύεται σαφώς ε, στην νομοθεσία υπάρχει ε, μία σαφής παραβίαση της νομοθεσίας εάν κατατέμνει κανείς το πρόγραμμα και έτσι επεμβαίνει ή στην ε, φύση των Άλπαιων η οποία είναι πολύ ε, αισθητή και πρέπει να διατηρηθεί. Ευχαριστώ η ε, συνάδελφος Βέτνεμαν. Και εγώ συμφωνώ με την προλαλή σας και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες με εντυπωσίασαν κατά την ανάγνωση αυτής της εκθέσεως διότι εδώ μιλάμε ε, για την δημιουργία ενός, ε, μιας λίμνης αποθηκεύσεως νερού και φαντάζομαι ότι και αυτό αναφέρεται σε ορισμένα εκτάρια που πρέπει να συνυπολογιστούν. Τώρα, ε, αν δεν λαμβάνει κανείς υπόψη τους επόμενους αναβαστήρες και δεν τους συνυπολογίζει είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω διότι ε, με την ίδια λογική θα μπορούσε κανείς να περιορίσει τις, τους χώρους στραθμέσεως. Ε, στην περιοχή που μένω εγώ παλιά υπήρχε ένα χωριό όπου υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πλέον ούτε ένα εκτάριο έδαφος και αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως ε, εξήγησε η συνάδελφος στην οδηγία ΕΠΕ υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις και εδώ μιλάμε για την κατάσταση του 2007 όπου πολύ συνειδητά υπήρξε σαλαμοποίηση, υπήρξε αφαίρεση ορισμένων συστατικών στοιχείων και το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Το άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ο τουρισμός μειώνεται και αναρωτιέμαι κατά πόσον χρειάζεται αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο ακόμη και είναι επίκαιρο επίσης υπάρχει μία γεωλογική αξιολόγηση που θεωρείται αντιεπιστημονική είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι μία γεωλογική αξιολόγηση είναι αντιεπιστημονική πώς απαντάει κανείς σε αυτή την περίπτωση Κύριο Ποστινάρου, Πάλι έχουμε εδώ πέρα déjà vu. Και εγώ κάτι αντίστοιχο το έχω ζήσει στη δική μου χώρα. Υπάρχουν διάφορα επιτίδη που προσπαθούν να παρακάμψουν το νόμο και ουσιαστικά σαλαμοποιούν το πρόγραμμα σε διάφορα κομμάτια. Ε, κάθε τμήμα υποτίθεται ότι είναι, σέβεται ας πούμε τα όρια, οπομένως περνάει. Αλλά όμως αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σφαιρικά. Δεν πρέπει να εξετάσουμε μόνο, δεν πρέπει να εξετάσουμε κάθε τμήμα του προγράμματος χωριστά. Και διερωτώ με γιατί η Κομισιόν δεν εξέτασε αυτά τα προγράμματα ε, με τρόπο σφαιρικό. Περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορείτε να σχεδιάσετε τα πάρκινγκ ε, χωριστά, τις πίστες χωριστά. Όλο το πρόγραμμα οικονομικός πώς και κοινωνικός πώς ε, είναι ένα πράγμα. Και αυτό είναι σαφές. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδεί τα συμπεράσματά της και τις απόψεις της και να επανέλθει στην Επιτροπή και να μας πει κατά πόσον υπάρχει πλήρως, ε, πλήρη σεβασμός της ε, οδηγίας και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο κύριος Βίλαντ. Ναι. Τώρα όμως πρέπει να διορθώσω διάφορα θέματα, διότι επανέρχομαι στο χώρο σταθμεύσεως που ήταν προϋπάρχον χρησιμοποιείτο, χρησιμοποιείτο ελάχιστα και τώρα χρησιμοποιείται περισσότερο. Δηλαδή ε, αυτό ισχύει για το χώρο σταθμεύσεως, το πάρκινγκ. Αλλά ε, όσον αφορά την λίμνη για το τεχνητικό χιόνι, ε, μας είπαν ότι χρησιμοποιήσανε μία παλιά λίμνη που υπήρχε για τεχνητό χιόνι για το νέο για το νέο χιονοδρομικό. Δηλαδή δεν υπάρχει μία τακτική σαλαμοποίησεως αλλά αυτό που ελέγχθηκε είναι σωστό είναι ότι πρέπει να αξιολογήσουμε το συνολικό πρόγραμμα και να δούμε και πέρα το ορίζοντα της πενταετίας διότι ε, υπάρχει μία σκόπιμη, μια σκόπιμη διατύπωση η οποία υπευλήθη και θα πρέπει ε, σε ένα άλλο χρονικό σημείο να δούμε εάν ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο μπορεί ε, και θέλει να προσφέρει ε, εμπόδια και αν θέλουμε να υπάρξουν αυτά τα εμπόδια. Λοιπόν, αναφέρομαι καταρχήν στη σαλαμοποίηση και δεύτερον εις, ε, την, ε, στην παραγωγή τεχνητού χιονιού για συγκεκριμένες πίστες και στην αξιολόγηση εάν οι αυστριακές αρχές έχουν εφαρμόσει νομοθεσία σωστά. Δεν νομίζω ότι οι σκοπίμως οι αρχές έκαναν κάτι παραπάνω από ό,τι επιτρεπόταν. Ευχαριστώ. Προφανώς πρέπει να επανέλθουμε και να ξανασυζητήσουμε το σημείο αυτό. Ο κύριος Βίλαντ θα αξιολογήσει εάν χρειάζεται κάτι παραπάνω πριν ψηφίσουμε το τελικό έγγραφο, το οποίο μας έχει ήδη παρουσιάσει υπό την πρώτη του μορφή. Κυρία Πρόεδρε, η πρότασή μου ήταν να αλλάξουμε τη μορφή και τώρα να διοχετεύσουμε το όλο θέμα μέσω μίας προφορικής ερωτήσεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσουμε μία απάντηση από τον Επίτροπο και μετά να δούμε αν ε, θα χρειαστεί μία αλλαγή της οδηγίας ΕΠΕ επί του συγκεκριμένου θέματος. Για την πρόταση Δίλαντα. Νομίζω ότι είμαστε σύμφωνοι, υπάρχει ομοφωνία. Φυσικά θα μιλήσουμε στη συνάντηση των συντονιστών και θα δούμε ποια είναι η καταλληλότερη στιγμή για να το συζητήσουμε και θα ζητήσουμε από τον κύριο Βίλαντ να αλλάξει το κείμενο για να συζητούμε επί ενός ολοκληρωμένου και διαμορφωμένου εγγράφου. Ευχαριστώ τους αναφέροντες. Θέλετε να απαντήσετε. Η συζήτηση, κοιτάξτε, δεν έχει κλείσει. Θα παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ένα λεπτό σας δίνω. Πολύ σύντομα θέλω να προσθέσω κάτι. Πολλοί εμπειρογνώμονες στην περιοχή θεωρούν ε, την περιοχή Ραγκάτσερ Πλάνκεν ε, ότι σαν μια περιοχή φυσικού κάλους που δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Ε, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι έχουν υπάρξει σημαντικές επιδεινώσεις και ένα βασικό μέρος της, όπου διαβιούσαν διάφορα θυράματα έχει καταστραφεί. Θα έπρεπε λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση να εξεραταστεί και ε, να ελεγχθεί. Ευχαριστώ. Παίρναμε στην αναφορά 20. Ο David Petri ε, είναι αναφέρον και έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Για επί 20 χρόνια η Ιταλία ε, αντιμετωπίζει με διακριτικό τρόπο τους μη Ιταλούς το Ιταλικό καθηγητικό προσωπικό σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη θέση απασχόλησης, τη διάρκεια των συμβολέων, την ίση ε, αμοιβή και τα στεξιωτικά δικαιώματα. Και το δικαστήριο έχει αποφασίσει υπέρ των λεκτών έξι φορέ. Όλοι γνωρίζουμε ότι πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εισήγαγαν ε, νομοθεσία που πολύ συγκεκριμένα αφορούσε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, ε, τους αφαίρεσε τα αστικά του δικαιώματα, του κατέστησε ξένου και εν πάση περιπτώσει όχι ε, νομικά πρόσωπα, οι φυσικά πρόσωπα που έχουν τα ίδια δικαιώματα ε, με τους υπόλοιπους ε, πολίτες. Από την πρώτη υπογραφή της ε, συνθήκης στη Ρώμη το 1957 μέχρι τη συνθήκη της Λισαβόνας, πολλές κυβερνήσεις, κάποιες περισσότερο από άλλες, παραβίασαν τις συνθήκες που είχαν υπογράψει. Παρ' όλα αυτά, δεν γνωρίζω καμία κυβέρνηση που προσυπέγραψε αυτές τις συνθήκες, η οποία έχει νομοθετήσει ενάντια στις συνθήκες και στην εξουσία του 10. Ε, ορισμένοι από, εσάς μπορεί να φαντάσετε ότι αυτό είναι απίστευτο. Στην πραγματικότητα όμως είναι λιγότερο από 100 ώρες μακριά από μας. Ε, το Σάββατο αυτή τη βδομάδα, 29 Ιανουαρίου 2011, ένα ιταλικό νόμο, η μεταρρύθμιση Τζελμίνη, ε, τέθηκε σε ισχύ και μου αφαίρεσε και εμένα και σε άλλου ε, συναδέλφου βασικά αστικά δικαιώματα. Από το Σάββατο το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση δεν υπάρχει. Το απαραβίαστο δικαίωμα τη υπεράσπιση. Δεν υπάρχει. Το δικαίωμα στην, στα ένδικα μέσα. Δεν υπάρχει. Το δικαίωμα ε, να υπάρξει απόφαση από δικαστή ε, σε τα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει. Ακυρώθηκε από το άρθρο 26 του νόμου Τζελμίνη. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Τζόρτζο Ναπολιτάνο, ε, παρότι υπέγραψε το νόμο αυτό, ανέφερε το άρθρο 26 ως ένα άρθρο προβληματικό, το οποίο θα πρέπει να επανεξεταστεί. Αυτό που δεν έκαναν ποτέ οι Ρωμαίοι, το έκανε μια Ιταλική κυβέρνηση. Πώς στάσαμε σε αυτό το σημείο και γιατί. Γιατί το Ιταλικό κράτος έλαβε τέτοια δραστικά μέτρα. Η απάντηση. Για περίπου 20 χρόνια τα πανεπιστήμια σε όλη την Ιταλία ε, έχουν δαπανίσει εκατομμύρια ε, λόγω του ότι έχουν γίνει ε, αγωγές από ξένους, ξένο διδακτικό προσωπικό για θέματα ίσης αμοιβή. Υπάρχουν εκατοντάδες ε, δικαστικές υποθέσεις εκκρεμής. Ε, και παρά το αργό νομικό σύστημα της Ιταλίας, στην πραγματικότητα βρίσκεται λύση αργά-αργά. Το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, παραδείγματο χάρη, ε, διατάχθηκε να πληρώσει 5 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις γιατί καθυστέρησε να πληρώσει διάφορους μισθούς σε 14 λέκτορες. Ε, τα πανεπιστήμια λένε όμως ότι έχουμε χρεοκοπήσει, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, το κράτος λέει δεν θα πληρώσουμε. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε, δεν θα πληρώσουμε. Η κυβέρνηση του Μπερλουσκόνη ε, βρήκε την εξή λύση. Είναι να εξαλείψει τις αγωγές των λεκτόρων. Αυτό λέει το άρθρο 26. Καταργεί όλες αυτές τις εκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Ε, νομοθετώντας λοιπόν εναντίον των αποφάσεων του ΔΕΚ και νομοθετώντας εναντίον των ευρωπαϊκών συνθήκων μας αφαιρεί, τα πλήρη δικαιώματα που έχουμε ως πολίτες. Χθες οι δικηγόροι μας έγραψαν στην Κομισιόν και ζήτησαν διαδικασίες επί παραβάση. Ζητάμε από την Επιτροπή σας να ζητήσει την γρήγορη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητήσει να εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών το θέμα και να ζητήσει από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου να συγγράψει την έκθεση για αυτό το θέμα, δεδομένου τη σοβαρότητα τη αναφορά μα. Και ζητάμε από την Επιτροπή να αναφορά να κάνει μια δημόσια δήλωση στα ΜΜΕ. Ζητάμε αυτή η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα θεμελιώδη νομικά μα δικαιώματα, ε, εμά των μη Ιταλών πολιτών, να αποκατασταθούν στην δημοκρατία τη Ιταλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ε, Δημήτριος Κοντιζάς. Ah, oui. merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ. Μας απασχολεί αυτή η υπόθεση εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Υπήρξαν διαδοχικές αποφάσεις του 10 που επιβεβαίωσαν ότι η Ιταλία δεν σεβάστηκε τις υποχρεώσεις της με βάση τη συνθήκη και κυρίως του άρθρου 45 για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, μια και οι ξένοι κθένης υπηκότητας λέκτορες ε, τη χάνουν ε, μεταχειρήσεων σε σχέση με τους Ιταλούς. Ε, στις 17 Ιουλίου 2006 το 10 αποφάσισε παρά την αντίθετη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι με βάση το νόμο 63 του 2004 υπήρχε επαρκές νομικό πλαίσιο για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των λεκτόρων, των παλαιών λεκτόρων ε, ξένων γλωσσών, που με τη μεταρρύθμιση του 1995 έγιναν συνεργάτες και ειδικοί εμπειρογνώμονες για θέματα γλωσσών. Είμαστε σε μόνιμη επαφή με τους αναφέροντες και την ε, οργάνωση που τους εκπροσωπεί και είμαστε δεστοποιημένοι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι λέκτορες ξένων γλωσσών. Το, το... Η απόφαση του 10 του 2006 μας έδαινε τα χέρια. Γιατί αν εκινήτω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει υπόψη της ε, γεγονότα που αφορούν ε, ή μάλλον δράσεις του Ιταλικού κράτους. Μιλάμε για κακή νομοθεσία ή κακές πρακτικές ό,τι αφορά το κοινοτικό δίκαιο. Κακές πρακτικές, δηλαδή διοικητικές πρακτικές, ε, που γίνονται κατ' εξακολούθηση και γενικής φύσεως. Το νομικό πλαίσιο πιστεύουμε ότι ήταν επαρκές ό,τι αφορά τις κακές διοικητικές πρακτικές. Είμαστε σε μόνιμη επαφή με την οργάνωση των λεκτόρων ξένων γλωσσών για να διαπιστώσουμε κατά πόσον υπάρχουν τέτοια προβλήματα κακών πρακτικών και να, για να μας γνωστοποιηθούν κακές πρακτικές ε, που δημιουργούν διακρίσεις. Τώρα, υπάρχει ένα νέο γεγονός το οποίο μόλις μάθαμε, η μεταρρύθμιση που αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Η Κομισιόν σε αυτή τη φάση περιμένει με μεγάλη προσοχή την εφαρμογή αυτής της νέας νομοθεσίας. Έχουμε αμφιβολίες για, την, για το σύμμορφο με το άρθρο ή μάλλον το σύμμορφο του άρθρου 26 της νέας νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο όπως το ερμήνευσε το ΔΕΚ για την κατάσταση των λεκτόρων. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω και διαβεβαιώνω και τους αναφέροντες που είναι λέκτορες ότι η Κομισιό θα κάνει ό,τι μπορεί και θα ξεκινήσει αν χρειαστεί τις απαραίτητες διαδικασίες αν διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα δηλαδή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. sorry. Just, uh, just, uh, Θέλω να υποστηρίξω την ε, αναφορά. Ότι δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε κάποια κίνηση, κάποια δήλωση εμεί από πλευρά τη Επιτροπή μα, διότι νομίζω ότι αυτά είναι πάγια προβλήματα. Οπότε και εγώ έρχομαι να συμφωνήσω με την πρόταση. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Είναι μια οριακή περίπτωση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Αναφορών Εδώ και πάνω από 15 χρόνια έχουν εξετάσει το θέμα. Ο χρόνος είναι απίστευτα μακρύς, ε, η προθεσμία δηλαδή. Ε, το δικαστήριο έχει λάβει καταδικαστικές αποφάσεις. Ε, έχει ασχοληθεί κατά επανάληψη με το θέμα αυτό. Η ιστορία αυτή μας κάνει να πρέπει να σκεφτούμε για τα μέσα και τις εγγυήσεις που προσφέρουμε στους πολίτες. έστω και μέσω της Επιτροπής Αναφορών, της οποίας είμαι πρόεδρος. Αυτά που είπε η κυρία Όκεν θα πρέπει να σε απασχολήσουν πιο ευρέως. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Παρότι δεν το λέω ρητός, νομίζω ότι συνειδητοποιώ ότι η νέα νομοθεσία που ενέκρινε το Ιταλικό Κοινοβούλιο και που ανέφερε αναφέροντας την παρουσίασή του, έχει ένα τέτοιο περιεχόμενο που μπορεί να έχει νόημα να στραφούμε προς το δικαστήριο για να επανεξετάσει την υπόθεση. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει μέχρι στιγμή. σω είναι λοιπόν αυτό το στοιχείο, αυτό το, καινο, το, το καινοτόμο στοιχείο, για να ζητήσουμε μία διαδικασία αναθεώρηση από το δικαστήριο. Περιμένουμε την αξιολόγηση τη ε, Κομισιόν για τον νέο νόμο και ακριβώ μέχρι ε, τότε θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Επίσης, μπορούμε να στραφούμε προς τις τελικές αρχές. Για να καταλάβουμε, πέρα από την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που υπάρχει. Θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε να έρθουν εδώ στην Επιτροπή μας, ας πούμε για να μας παρουσιάσουν με σαφή τρόπο το πνεύμα αυτού του νέου νόμου και κατά πόσο είναι σύμμορφο με το άρθρο 26. Θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν την άποψη της Ιταλικής κυβέρνησης για αυτό το παλιό πρόβλημα της Ιταλίας. <laughs> Αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά λοιπόν και ελπίζουμε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα οι Ιταλικές αρχές. Ο κύριος Γιάρ. Καταρχήν συμφωνώ απολύτως με την πρόταση της Προέδρου και δεύτερον δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν πιστεύω ότι έχει δυνατότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι τόσο αδύναμη και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, τότε μπορεί βάσει της ε, συνθήκης ε, ε, κάτι να κάνει. Δηλαδή μπορεί να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις. Δηλαδή αυτό πρέπει να διαπιστώσουμε είναι αν είναι σωστό ή όχι. Αλλά θέλω να συμπληρώσω στην πρόταση της Προέδρου ότι θα ήθελα την ε, ε, ε, αναφορά αυτή να την επανεξετάσουμε εντός του έτους και όχι να περιμένουμε εσαΐ. E. Δηλαδή κάτι να γίνει και αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι πάλι κάτι θα πρέπει να γίνει. Θα ήθελα λοιπόν συντόμως να ξαναδώ αυτό το θέμα στη συνεδρίασή μας. Ο κύριος, Μποστινάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ τώρα νιώθω έκπληξη. Τι είναι αυτό εδώ, αυτό είναι η αναβολή στις ρωμαϊκές καλένδες ή είναι κάτι σαν πιστοποιητικό θανάτου. Τι, μα τι, τι γίνεται εδώ πέρα. Για να λύσετε το πρόβλημα, κύριε και κυρίες επιτροπές, πρέπει να κάτσετε να κρίνετε εάν υπάρχει εδώ παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Μπορείτε να μας απαντήσετε ευθέω. Όχι από ό,τι φαίνεται. Κάτι άλλο. Εδώ πέρα κυρία Πρόεδρε, ε, έχουμε μια περίπτωση που παρομοιάζει με εκείνη που αφορούσε την Αγγλία, το Βρετανικό Δίκαιο, όπου δεν αναγνωρίζουν σε έναν φαρμακοποιό Γάλλο να ανοίξει φαρμακείο στο Εμένο Βασίλειο. Σήμερα, επομένως, έχουμε άλλη μια τέτοια περίπτωση, ένα κράτος μέλος να απαγορεύει σε ένα ξένο ε, πανεπιστημιακό να πάει και να διδάξει σε ένα πανεπιστήμιο στη χώρα την εν λόγω. Εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να λύνει τέτοια προβλήματα. Αλλιώς παραβιάζεται την συνθήκη της Λισαβόνας. Παίζεται με τα σύμβολα. Πολύ κομψό, αλλά παράδειγμα. Ε, Ευχαριστώ. Ο αναφέρον για ένα λεπτό. Σε περίπτωση που θέλει να προσθέσει κάτι. Ε, Απλώς πρέπει το λόγο να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε φέτος. Ευχαριστώ. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την αναφορά που αναφέρεται στο σημείο 21. Ο αναφέρον έχει το λόγο. Muito Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους, λέει. Ο υποβάλλοντα την αναφορά γιατί θέλω να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα για την ευκαιρία μου δίνετε που με καλέσατε και επίσης έτσι ε, δεν έχουμε απλώς ένα τέτοιο έργο το οποίο αφορά τις τουριστικές ΜΜΕ. Παρά από αυτό εδώ έχουμε κάποιες βασικές ε, ε συνθήκες που διέπουν την αγορά και τις ε, και, το, και τον κλάδο αυτό όσον αφορά κάποιες ε, ε, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην Πορτογαλία. Γι' αυτό και θέλω να σας επισημάνω ε, ότι εδώ πέρα έχουμε μία ευρωπαϊκή απόφαση και θέση που δεν καταλαβαίνω θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ε, ευθύς εξ αρχής σας λέμε ότι έχουμε το, τον Νοέμβριο 2008 κάποιες υποψηφιότητες και αυτό ε, είχε γίνει τότε με κάποια καθυστέρηση. Θα έπρεπε επομένως να υποβάλουμε συμμετοχή στον διαγωνισμό με δύο χωριστές αιτήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έλαβε από εμάς ε, όλη την τεκμηρίωση και προέκυψε ότι υπάρχει εδώ πέρα ασυμβατότητα ε, ότι υπάρχει επίσης και απουσία νομιμοποίησης. Οπότε, στη συνέχεια είχαμε τροποποίηση του πορτογαλικού δικαίου, ζητήθηκαν επομένως το 2009 παραπάνω πληροφορίες. Πρόκειψε και πάλι ότι σε σχέση με το άρθρο 19 παραγωγός Β είναι ε, πάλι απαράδεκτη αυτή η αίτηση. Αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες ε, ε, μέσω κάποιας ε, χρηματοδότησης θεωρούνται ως εταιρείε εμπορικές οι οποίες μπορούν να κάνουν αυτού του είδους τις καμπάνιες και έτσι να προάγουν τον τουρισμό στο ιστορικό και στο εξωτερικό. Ο δικό μας φορέας ισχυρίζεται ότι ο ανώτατος φορέας ήταν και είναι ένας τέτοιος τεχνικός οργανισμός και αυτή η κρέν, αυτό, αυτός ο φορέας, θεωρούμε ότι μας έχει προκαλέσει ζημία. Ε, αρχές Δεκεμβρίου 2010 διαβιβάσαμε αρμοδίως και άλλη τεκμηρίωση και έτσι προσπαθούμε να καταδείξουμε ότι υπάρχει παραβίαση προηγουμένης συμφωνίας του 2008. Αυτή η τεχνική οργανισμή του ΚΡΕΝ μας ε, υποχρέωσαν με κάποιες ε, αποφάσεις παράνομες και καθυστερημένες ε, επί εννέα μήνες να ασχοληθούμε με αυτή την περίπτωση και έτσι καθυστέρησε η αναδοχή του έργου. Επίσης, οι τεχνικοί οργανισμοί της ΚΡΕΝ αλλά και η κυβέρνηση της χώρας ε, μας οδήγησαν σε κάποια σύγχυση σε σχέση με το ποιο, είναι αρμόδιος για αυτές τις ε, Και αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν αυτούς τους κανονισμούς μας οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Το 2004 άρχισα εγώ να ασχολούμαι με αυτόν τον κλάδο και ήλπιζα ότι θα βοηθηθώ από, τις, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γιατί αυτές οι αποφάσεις πρωτογενής δικαιοσύνης μας δημιούργησαν υλικές ζημίες, μας προκάλεσαν και επίσης ηθική βλάβη. πρόκειται για στρέβλωση της λογικής. Αυτό δεν είναι το ευρωπαϊκό οικονομικό πρότυπο. Τον Ιούλιο του 2009 και μετά επίσης ε, ενημερώσαμε τις ευρωπαϊκές αρχές, ε, ακολούθησε η νομοθεσία του 2011 που προέβλεπε δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθηθούν αυτές οι δράσεις. Και θεωρούμε ότι η οικονομική και η κοινωνική συνοχή της Πορτογαλίας δεν θα επιτευχθεί εάν παρεμποδίζονται με τέτοιες ενέργειες οι πορτογαλικές επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν φυσικά να δίνονται κίνητρα για ενέργειες καταχρηστικές αθέμητων ανταγωνισμού. Ουσιαστικά το, το δημόσιο ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και ε, απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατεπηγόντω να ασχοληθεί και να λάβει υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα. Επίσης θα πρέπει οι πορτογαλικές αρχές να πάψουν να εφαρμόζουν αυτήν την στρεβλή λογική. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Κομισιόνα Dirk Peters. Dirk Peters από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, έχω ήδη επαφή με τον ε, αναφέροντα για να τον γνωρίζω. Ε, στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για δημόσιους διαγωνισμούς για περιοχές συγκλήσεως στην Πορτογαλία που στηρίζονται από επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το θέμα αυτό αναφέρεται στην ε, πολιτική συνοχής και στα διαρθρωτικά ταμεία που εφαρμόζονται μέσω της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπου δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει εις, ε, δεν συμμετέχει άμεσα στην επιλογή των εκατοντάδων προγραμμάτων. Αυτό είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να φροντίσει ώστε οι εθνικές αρχές στην επιλογή των προγραμμάτων να προχωρήσουν βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας. Γι' αυτό και ελέγξαμε διεξοδικά τα στοιχεία που μας ε, υποβλήθηκαν και στις αρχές ε, του Μαΐου στείλαμε ένα εκτενές ερωτηματολόγιο στις ε, πορτογαλικές αρχές που μας απαντήθηκε τέλη Ιουνίου και το οποίο αναλύσαμε και σε πολλά σημεία οι απαντήσεις αυτές δεν μας ικανοποίησαν. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγο πριν τα Χριστούγεννα απίφθινε με ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο στις πορτογαλικές αρχές με 13 σελίδες λεπτομερών ερωτήσεων και η απόφαση αυτή μας, ε, μας την έχουν υποσχεθεί για την Παρασκευή αυτής της εβδομάδος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσετέθηκε άλλη μία πτυχή ε, σχετικά με αυτή την νομοθεσία η οποία δίδει μία ιδιαίτερη θέση εις ε, την Διεύθυνση Επενδύσεων της Τουρίσμο de Portugal όπου ζητήσαμε να μας διευκρινίσουν εάν αυτός ο κρατικός οργανισμός μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω διαρθρωτικών πιστώσεων για προγράμματα τα οποία οργανώζουν ιδιώτες αναδοχή όπως η εταιρεία του κυρίου Μάτους. Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε αν πρέπει να εμπλέξουμε και την περιφερειακή περιοχή. Δηλαδή εάν ε, υπάρχει συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής ε, της ε, διεύθυνσης αυτής και αυτό είναι θέμα εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά πρέπει να δούμε εάν οι πιστώσεις ενός δημοσίου οργανισμού συνάδουν να χρησιμοποιούνται και σύμφωνα με το ιδιωτικό δίκαιο. Όπως σας είπα, η απάντηση αναμένεται για την Παρασκευή. Στην ε, πρώτη ε, απάντηση ε, μας ελέγχθη ότι δεν είχε υπάρξει πλήρη εξήγηση του πόσο χρησιμοποιούνται οι πιστώσεις αυτές. Δεν μας είπαν ποιος ήταν ο τελικός αποδέκτης. Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί τώρα και ο ετών ε, ε, μάλλον ε, μία μία εταιρεία η οποία προωθεί την απάντηση ενός ιδιώτη και πρέπει να αιτιολογήσει αν η διαδικασία της απονομής του διαγωνισμού ήταν σωστή ή όχι ο κύριος Γιάρ. Αλλά ουσιαστικά τελειώνουμε κύριε Γιάρ. Δηλαδή, εάν κατάλαβα καλά, τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχουν ακόμη όλες οι πλήρεις πληροφορίες άρα πρέπει να διαθέσουμε τον αναγκαίο χρόνο προτού λάβουμε την τελική απόφαση πολύ γρήγορα. Καταρχάς να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Δεύτερον, να περιμένουμε την τελική απάντηση της πορτογαλικής κυβέρνησης και να κρίνουμε με τα λόγου γνώσεως. Ε, εντάξει, περιμένουμε λοιπόν την απάντηση λέει πρόεδρος των πορτογαλικών αρχών. Ο αναφέροντας, αλλά πολύ σύντομα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους αξιούς βουλευτές διότι με καλέσατε εδώ και θέλω να τονίσω το ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση αυτής της ε, διαδικασίας κατά την οποία αφού εχρησιμοποίησαν της κυβέρνησης τους πόρους του Διαρκτικού Ταμείου με τρόπο παράλογο είναι τώρα το πιο σημαντικό να εξασφαλιστεί το δίκαιο και αίσιο πέρας αυτού του σύριαλ. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα διότι μιλούμε για εμάς που είμαστε θύματα δημοσίας επιθέσεως. Έτσι μας αποθαρρύνουν, έτσι μας απομονώνουν και δεν μπορούμε έτσι να ασκήσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Ωραία, αφήνουμε ανοιχτή αυτή τη φορά. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι έλαβα δύο αιτήματα από την Τατιάνα Ζανόφσκα να περάσει μια αναφορά από το σημείο Β στο σημείο Α, από την κυρία Όκεν την αναφορά να περάσουμε την αναφορά επίσης από τη 1772-2009 και επίσης να κάνουμε ένα ερώτημα προς την Επιτροπή Αλίας και την Επιτροπή ΙΜΚΟ, χωρίς όμως να ανοίξουμε αυτή την αναφορά, χωρίς να την περάσουμε στο σημείο Α. Ευχαριστώ. Κλείνω εδώ οι εργασίες της Επιτροπής μας.